Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Καταρχήν, να σας προειδοποιήσω ότι θα έχουμε web streaming της συνεδρίασης ε, και θα υπάρξει και ματογράφηση. Σήμερα θα συζητήσουμε τις θεσμικέ πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, σύμβαση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδες Ελευθερίες. Βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή, γιατί η πρόκληση που θέτει η Συνθήκη της Λισαβόνας συμπεριλαμβάνει και την πτυχή αυτή, που Καταρχήν αφορά τη δική μας επιτροπή. Υπάρχει ήδη νομική υποχρέωση για την προσχώρηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αν και υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θέλουμε σήμερα να τα συζητήσουμε μέσω αυτής της ακρόασης με ένα ξεκάθαρο τρόπο για να αποφύγουμε να υπάρχουν στη συνέχεια δυσκολίες ή επιπλοκές στη στιγμή της κύρωσης της συνθήκης. Έχουμε ήδη συζητήσει στην Επιτροπή μας ε, και ε, είχαμε επίσης και συζήτηση και στην Επιτροπή για τις ε, ελευθερίες. Οι εργασίες της σχετίζονται με τις εργασίες της δικές μας Επιτροπής. Έτσι λοιπόν συζητήσαμε τα θέματα αυτά και υπήρξε και ο συνάδελφος Χαρέγου, ο οποίος ε, εκπώνησε τη σχετική έκθεση. Είχαμε και τη συνάδελφο Γκάλ από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Χαιρετίζω όλους τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται εδώ και εκπροσωπούν ε, τους εθνικούς θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον ακαδημαϊκό τομέα θα πρέπει να ανακοινώσω ότι ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου των Κάτω Χωρών, ο κ. Βαντελίντεν, δεν θα έρθει, γιατί δυστυχώς ε, υπάρχει μια ανακρόσιμη ακολουθία του Υπουργού Εξωτερικών Χάνσεν Μέρλο και πρέπει να παρευρεθεί. Έτσι λοιπόν ε, θα ακολουθήσουμε την εξής πορεία της μας. Αρχικά θα έχουμε μία σύνοψη των σκέψεων και των συζητήσεων που είχαμε στην Επιτροπή αυτή από τον κύριο Ραμόν η Πρέπει να είστε σύντομος για να μπορέσουν όλοι να τοποθετηθούν. Όμως, ε, αν δεν ε, έρθει ο αξιότιμος συνάδελφος στα 15 λεπτά, θα Πρέπει να διακόψουμε κατόπιν. Η κυρία Κιγκαγκάλ ε, θα παρουσιάσει τη δική της έκθεση, εκπρόσωπος της Επιτροπής ΛΥΠΕ και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονε μας και φυσικά θα υπάρξουν και ρωταπαντήσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Χαρέγκουι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω θα μπορέσω να συμμορφωθώ προς τα υποδείξει σας σε σχέση με τον χρόνο ομιλίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες για την παρουσία τους. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα σήμερα και ιδίως με μεγάλο ενδιαφέρον γιατί η έκθεση αυτή που αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πέραν από την απλή πολιτική και νομική απόφαση που εμπεριέχει έχει και μια πάρα πολύ σημαντική τεχνική πολυπλοκότητα. Η ιδέα λοιπόν του να οργανώσουμε, να διοργανώσουμε αυτή την ακρόαση με πολλούς πάνω από μια ντουζίνα εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά, είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να δώσει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και θα εμπλουτίσει τη συζήτησή μας σε τεχνικό επίπεδο και θα μας ε, βοηθήσει, ελπίζω, να επιλύσουμε πολλά ερωτηματικά, πολλά στοιχεία που είναι άγνωστα και αστάθμητα για πολλές πτυχές οι οποίες συνάπτονται με την προσχώρηση της σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χθε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας πληροφορήσω για αυτό. Χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εντολή διαπραγμάτευση για την προσχώρηση στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η είδηση και πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε την ευκαιρία σε άμεσο χρονικό διάστημα να θέσουμε αυτό το ερώτημα στην κυρία Ρέντινγκ, η οποία θα εμφανιστεί λίγο αργότερα στη συνεδρίασή μας, σε σχέση με τις παραμέτρους που καθορίζουν αυτή την εντολή διαπραγμάτευσης. Γιατί από χθε, με τρόπο επίσημο πια, ξεκινά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η εντολή ώστε να υπάρξει πλήρης προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Προφανώς αυτή η εντολή στη συνέχεια θα πρέπει να τύχει ομόφωνη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα ή μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Και πιστεύω ότι αν δεν υπάρξουν δυσκολίες, αλλά πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες γιατί ορισμένε χώρες μπορούν να θέσουν αντιρρήσεις και προσκόμματα από ό,τι γνωρίζω. Αν μπορέσουν όμως να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα, μπορούμε να προβλέψουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει την εντολή αυτή διαπραγμάτευσης ομόφωνα μέσα στους επερχόμενους μήνες, ακόμα και μέσα στις επερχόμενες εβδομάδες, το ελπίζω. Και από εκεί και πέρα μπορεί να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Τώρα με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ίσως και το αντικείμενο της σημερινής ημερίδας σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα καταρχήν να κάνω μία απαρίθμηση και κατάταξη των ερωτηματικών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα πρώτο ερώτημα αφορά το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί στη συνέχεια με τις παρεμβάσεις των διαφόρων εμπειρογνωμών θα αντιμετωπίσουμε πολλά θέματα, πολλά θέματα που όπως και θα αναφέρει και η κυρία Κίνγκα Γκάλ, εξ ονόματος Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, Υπάρχουν και άλλε επιτροπέ, όπω η Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων επίση που έχουν εκφράσει την άποψή του, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτή. Όλε οι επιτροπέ αυτέ λοιπόν θα προσφέρουν τη δική του συνεισφορά στα θέματα τη διαπραγμάτευση. Επομένω, το πρώτο θέμα είναι τα θέματα τη διαπραγμάτευση. Ποιο διαπραγματεύεται εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο εξ ονόματο τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Έχουμε 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα συμμετάσχουν όλα αυτά τα μέλη. Στη διαπραγμάτευση θα πρέπει να δώσουν την επιφόρτιση σε κάποιο. Και η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται σαν να ήταν ένα κράτος παραπάνω στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αλλά στην περίπτωση αυτή πώς θα γίνει σεβαστή η ιδιαιτερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι δεν είναι δηλαδή ένα κράτος, αλλά ουσιαστικά ένα σύνολο από κράτη, μια οργάνωση κρατών. Στη συνέχεια, <clears throat> ξέρουμε ποιες είναι οι εκθέσεις των άλλων επιτροπών και υπάρχει η διεκδίκηση όλα τα πρωτόκολλα και, το, και η σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι όλα αντικείμενο τη προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν πώ υπογράψει όλα τα πρωτόκολλα τα οποία προσαρτούνται στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κοινό παρονομαστή ε, για τα θέματα αυτά των πρωτοκόλων περιορίζεται μόνο σε δύο πρωτόκολλα. Άλλο ερώτημα. Πώς περιορίζεται η διαπραγμάτευση από το γεγονός ότι η συνταγματική εντολή της ε, συνθήκης της Λισαβόνας λέει ότι δεν θα πρέπει να ανατραπεί προηγούμενη νομική, το προηγούμενο νομικό καθεστώς των κρατών μελών. Άλλο ερώτημα. Είναι απαραίτητο, είναι πρόσφορο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει και σε άλλες συμβάσεις και πώς μπορεί να το πράξει χωρίς να ανατρέψει την ουδετερότητα που επιβάλλει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια άλλη συζήτηση, η οποία ξεκίνησε επίση στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, αφορούσε τι διάφορε τροπολογίε, οι οποίε νομίζω ότι ενεκρίθηκαν, με στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει σε μια σειρά από φορεί και οργανισμού που έλκονται από τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά που δεν είναι οργανισμοί οι οποίοι αναφέρονται εκπεφρασμένα στο, στη σύμβαση αυτή. Παραδείγματο χάρη φορεί που αφορούν τον το να είπα, το εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Επιτροπή κατά των, βασανιστήριων και όλα αυτά. Είναι λοιπόν διάφοροι φορείς οι οποίοι βρισκόνται κατά κάποιο τρόπο κάτω από την αιγίδα, κάτω από την ομπρέλα του, της συμβασία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, όπως λέει μια τροπολογία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ποιες είναι οι τεχνικο-διοικητικές πτυχές επίσης αυτής της που θα πρέπει να επιληθούν, ξέρετε, παραδείγματος χάρη ότι η συνεισφορά των κρατών που συμμετέχουν σε αυτή τη σύμβαση γίνεται επί τη βάση του ΑΕΠ. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ήδη καταβάλουν ως μεμονωμένα κράτη-μέλη <clears throat> τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύμβαση. Επίσης, πώς θα επιλέξουμε τους δικαστές οι οποίοι θα πρέπει να συμμετέχουν. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πρώτερη ακρόαση όπως αυτή που κάνουμε για τους ε, επιτρόπους για την επιλογή των δικαστών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 255 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη συζήτησή μας. Ποιος θα εκπροσωπεί επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσουμε. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούν να προσφεύγουν εναντίον άλλων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, γιατί αυτό είναι απαραίτητο αν λάβουμε υπόψη το άρθρο 344 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτεί την χρήση <clears throat> διαιτητικών μηχανισμών προτού υπάρξει κάποια προσφυγή ενός κρατούς μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός κάποιου άλλου. Πώς θα πρέπει να περιορίσουμε την πρόσβαση στο δικαστήριο του Στρασβούργου με προηγούμενες διαδικασίες, με μια προηγούμενη διαδικασία εξέτασης προσφυγών ενώπιον των δικαστικών αρχών των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, η παθητική νομιμοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών, πώ θα πρέπει να οριοθετηθεί όταν υπάρχουν προσφυγέ κατά των για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αν αυτό θα πρέπει να αποτελεί λοιπόν αντικείμενο προσφυγή κατά των κρατών μελών ή κατά τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του να είναι συνδιάδικη η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεναγόμενη καλύτερα όταν υπάρχει μία ε, προσφυγή κατά ενός κράτους μέλους. Ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Θα πρέπει να επισημοποιηθεί κάποιο πρωτόκολλο που συνδέει αυτά τα δύο δικαστήρια. Και ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις διαδικασίες που είναι εν εξελίξει ήδη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί θέλω να σας, να σας καταδείξω πόσο πλούσιος είναι ο τεχνικός χαρακτήρας, αλλά και πόσο πολύπλοκος είναι ο τεχνικός χαρακτήρας των θεμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βόλφαν και τον κύριο Σιφάουρη για την ανεκτήμητη βοήθεια της, τους για την ε, διοργάνωση αυτών των ημεριδών και εσάς για την παρουσία σας και πάλι όπως είπα. Ευχαριστούμε κύριε Κερδίσαμε πέντε λεπτά από την ομιλία σας το λόγο στην συγκίτρια για γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ελευθεριών και για Γκάλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι θετικό που μας δώσετε τη δυνατότητα και την πρόσκληση να συμμετέχουμε σήμερα στη συζήτηση. Είχαμε δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών και Ιστορικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό. Και το κύριο ερώτημα ήταν ο πολίτης τι κερδίζει από αυτά, ποια είναι η προστιθέμενη αξία για τον πολίτη. Και αυτά θα πρέπει να τα τονίζουμε. Ποια θα είναι η απάντηση στα ερωτήματα αυτά. όταν μιλάμε για την προσχώρηση στη σύμβαση. Είναι μεγάλη επιτυχία πρώτον να έχουμε δεσμευτικό χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και μετά την προσχώρηση στη σύμβαση. Το πρωτόκολλο 14 στην σύμβαση επικυρώθηκε, άρα έχει στρωθεί ο δρόμος για προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει τμήματα αυτής της σύμβασης. Το νέο στοιχείο είναι είναι η προσχώρηση της Ένωσης ως νομική οντότητα στη σύμβαση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Πώς μια νέα νομική οντότητα μπορεί να συνεδριάζει στα πλαίσια αυτής της σύμβασης. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλης πολιτικής και νομικής σημασίας προκειμένου να δημιουργηθεί μια υπηρετική έκταση, ένας υπηρετική έκταση χώρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το γνώμη αυτό θα φέρει μια νέα δυναμική στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Όμως, πρέπει να τονίσουμε για τους πολίτες να υπογραμμίσουμε λέω το ότι θα συμβάλλει σε ένα πιο ε, συνεκτικό εσωτερικό νομικό σύστημα στην Ένωση και οι πολίτες θα έχουν επιπλέον μηχανισμού εφαρμογής των δικαιωμάτων τους. Βέβαια, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς θα λειτουργεί το σύστημα. γιατί πολλές προσδοκίες υπάρχουν, πολλές ιδέες κυκλοφορούν και αυτό το είπαμε στη χθεσινή μας συνεδρίαση, δηλαδή η διάδοση των πληροφοριών εκ μέρους της Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη για την προστιθέμενη αξία για τον πολίτη πρέπει να κυκλοφορήσει πώς θα λειτουργεί το σύστημα, πόσο πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτό Διαφορετικά θα δημιουργήσουμε φρούδες προσδοκίες. Στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα έχουμε μια πιο συνεπή νομολογία από εδώ και μπρος. Βέβαια, χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τα νομικά και πολιτικά σημεία και θέματα τα ανάφερε ο συνάδελφος. Και θα συζητηθούν φυσικά σε σχέση με τη σύμβαση. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να τονίσω ότι στις διαπραγματεύσεις αυτά τα νομικο-τεχνικο-θεσμικά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά να λάβουν σωστές απαντήσεις. Διαφορετικά θα δημιουργήσουμε σύγχυση και μπορεί να υπονομεύσουμε το ίδιο το εγχείρημα. Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά τα τεχνονομικά εμπόδια δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόσχημα για να δοθεί υπερβολική συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. και επειδή το θέμα τέθη στην Επιτροπή μας και η σύμβαση αυτή δεν αφορά μόνο τα θεσμικά όργανα της Ένωση, αφορά και τους πολίτες, θεωρούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να ζητηθεί, να του ζητηθεί η γνώμη του σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και τελειώνω επισημένοντας το ότι χρειαζόμαστε επαρκείς πληροφορίες και κατευθυντήρες γραμμές για τη χρήση αυτού του οργάνου ή του εργαλείου όταν θα έρθει η στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την κυρία Κιγκάλ και αρχίζει η ακρόαση. Θα συνοψίσω τηλεγραφικά τα θέματα. όροι, τεχνικοί για την προσχώρηση, επιπτώσεις της προσχώρησης, σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων. Πρώτος, ο, ο καθηγητής Χωσέ Πάστορ έχω από το Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσια της Μαδρίτης. Ευχαριστώ. Μικρό. Μικρό. C'è πρέπει να πατήσετε το κουμπάκι. Έλεγα ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω στην ακρόαση αυτού του κοινοβουλίου που αφορά το θέμα της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Ρώμης του 1950 και ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής για την πρόσκληση και θα ήθελα να συγχαρώ τον συμπατριώτη μου και τον εισηγητή, τον κύριο Χαουρέγγι, για το σχέδιο ε, ψηφίσματος που έχουμε ενώπιον μας. Το leitmotiv ε, της ομιλίας μου θα μπορούσε να, να, το εξή η μακρά πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ασφάλεια δικαίου και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί αν ε, πράγματι μέχρι το 1970 το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ουσιαστικά δίσταζε να δυσφαλίσει αυτή την ασφάλεια από εκείνη την ημερομηνία. Το ΔΕΚ ξεκινά μια πορεία στην ομολογία που καθορίζουν τα σχετικά κριτήρια, κριτήρια ή παραμέτρους που όπως είναι γνωστό η συνθήκη του Μάστρικ του 1952 ε, επιβεβαίωσε ότι, είχαν, ότι ήταν οι κύριες αρχές του κοινοτικού δικαίου έτσι όπως ε, ορίζεται στις εθνικές νομοθεσίες και στις αρχές που διέπουν τα διεθνή μέσα όπου ανήκουν τα κράτη-μέλη κυρίως στη συνθήκη της Ρώμης του 1950. Παρ' όλα αυτά, ε, πέρα από την αναμφισβήτητη πρόοδο που επέφερε η εφαρμογή αυτής της κανονιστικής παραμέτρου, η κύρια συνέστηση ήταν ότι οι κοινότητε δεν είχαν φτάσει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας δικαίου σε ένα τόσο σημαντικό σημείο και τόσο ευαίσθητο σημείο όπως η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα έλλειμμα που ε, αφορούσε όχι μόνο τον κατάλογο των δικαιωμάτων και ελευθεριών προς προστασία, αλλά και τον ορισμό και το συγκεκριμένο βεληνικές. Γινόταν λόγος για ε, μια προτεραιότητα προστασία. Επομένως, για να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα, άνοιγαν δύο οδοί λύσει. Η πρώτη ήταν η Σύμβαση τη Ρώμη του 1950 που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Η άλλη οδό συνιστόταν στην ε, δημιουργία ενό αυτόνομου μέσου αποκλειστικό για τι κοινότητε και πρέπει να πω ότι και οι δύο οδοί ε, κάποια στιγμή αποπεράθηκαν η πρώτη αυτή η οδός τη προσχώρηση Πρέπει να ξέρετε ότι το 1979 η Επιτροπή θέτει στο Συμβούλιο το θέμα και μόνο το Μάρτιο του 1994 ζητείται από το δικαστήριο μια συμβουλευτική γνώμη σχετικά με το ζήτημα αυτό. Η γνωμοδότηση εκδίδεται το Μάρτιο του 1996 και εκεί αναφέρεται ε, το συνταγματικό πελληνικές της προσχώρησης ε, και η αναγκαιότητα για να τροποποιηθούν οι συνθήκες στο πρωτογενές δίκαιο και έπρεπε να περιμένουμε τη θέση σε ισχύ της 1ης Δεκεμβρίου του 2009 τις συνθήκες της Λισαβόνας έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έχει αποκτήσει ήδη ε, νόμικη προσωπικότητα σε διεθνές επίπεδο, υποχρεούται να προσχωρήσει στη Σύμβαση της Ρώμης, ε, κάτι που επιφέρει τη σημαντική συνέπεια της αποδοχής ε, της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως προς το η δεύτερη οδό, δηλαδή τη δημιουργία ενό αποκλειστικά κοινοτικού μέσου, πρέπει να πω ότι φτάνει στο τέλος τη, στις του Συμβουλίου της Νικέα το Δεκέμβριο του 2000. Πρόκειται για τη διακήρυξη και όχι για την υιοθέτηση. Διακήρυξη από Επιτροπή Συμβούλιο και Κοινοβούλιο τη χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όμως δεν βρισκόμασταν ενώπιον ενός ε, μέσου το οποίο θα είχε δεσμευτικά νομικά αποτελέσματα, αλλά πρόκειτο για ένα κείμενο ηθικού και πολιτικού χαρακτήρα, αν και ήταν ε, αρκετά σημαντικό. Ο, σήμερα αυξήθηκε η σημασία αυτή γιατί μετά την ε, συμπερίληψή του στη συνθήκη της Λισαβόνας η χάρτα της νίκαιας είναι υποχρεωτικά, υποχρεωτική νομικά. Επομένως, μετά τη θέση σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009 ε, της Συνθήκης της Λισαβόνας ε, και όταν καθίσταται αποτελεσματική προσχώρηση ή όταν θα καταστεί αποτελεσματική προσχώρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει δύο σημαντικά δεσμευτικά μέσα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και επιπρόσθετα θα υπάρχουν δύο διεθνεί δικαιοδοσίε για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Έκανε ένα γιγάντιο βήμα. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καθώς από μια ανεπαρκή ασφάλεια δικαίου πέρασε σε μια πλήρη νομική ασφάλεια, μια πλήρη ασφάλεια δικαίου και ενισχυμένη. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να είναι ικανοποιημένοι λοιπόν αφού η μεγάλη πορεία που ξεκίνησε από το 10 το 1970 μπόρεσε να καταλήξει το 2009 στον επίτευξη του καλύτερου δυνατού στόχου και ε, αυτό αναγνωρίζεται στο σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε ενωπιών μας. Έχοντας φτάσει στο σημείο αυτό, νομίζω ότι σε σχέση με την ε, συμφωνία προσχώρησης που προβλέπεται στο πρόσθετο πρωτόκολλο, ε, στο 8ο προς το πρωτόκολλο Συνδική Σαββόνας, μπορούμε να κάνουμε κάποιες ε, σκέψεις επιλεκτικές και όχι εξαντλητικές σκέψεις σε σχέση με το θεσμικό ευρωπαϊκό συντέριασμα μεταξύ του ΔΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων που θα το ονομάσω Δικαστηρίο του Στρασβουργού για τα κύρια αυτά θέματα στα κύρια αυτά θέματα αναφέρεται η πρόταση ψηφίσματο αυτού του κοινοβουλίου που μα παρουσίασε ο κ. Ραμόν Χαουρέγγι προλίγο. Το πρώτο σημείο είναι να δούμε ποιο από τα δύο δικαστήρια του Λουξεμβούργου ή του Στρασβούργου θα είναι το κύριο δικαιοδοτικό όργανο και ποιο θα είναι το επικουρικό. Ε, δηλαδή, σε ποιο θα πρέπει πρώτα να προσφύγει το άτομο που θεωρείται θύμα παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του και μπορεί να δικαστεί η υπόθεση σε ε, ένα όργανο της Ένωσης. Η απάντηση δεν ε, έχει αμφιβολίες. Θα πρέπει καταρχήν ε, να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο του Λουξεμβούργο και αν εξαντληθούν τα ένδικα μέσα στη δικαιοδοσία αυτή, τότε θα πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Αυτό προκύπτει από την, αρχή, από την εφαρμογή μιας μεγάλης αρχής του Διεθνούς Δικαίου Δικαιωμάτων ε, της επικουρικότητας, ε, δηλαδή η αρχή αυτή διακηρύσει το κύριο χαρακτήρα των εθνικών ενδικών μέσων και την επικουρική φύση των διεθνών μηχανισμών. Εξού και ο κανόνας αρθρού 35 της Σύμβασης της Ρώμας που επιβάλλει την αναγκαιότητα να εξαντληθούν τα εσωτερικά ενδικά μέσα για να γίνει αποδεκτή μια ε, προσφυγή. Έτσι λοιπόν, καθώς ε, έχει μεταφερθεί στους δεσμούς της Ένωσης η άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων των κρατών, τους μεταφέρθηκε επίσης και ταυτόχρονα ο κύριος χαρακτήρας της άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων. Όπως ε, πολύ ορθά λέγεται σε αυτή την σειρά των ιδεών, στην πρόταση του κυρίου Χαουρέγγι, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου σε σχέση με το Δικαστήριο του Στρασβούργου θα έχει μια ανάλογη θέση με τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών φυσικά στη συνεννόηση ότι σε αυτά τα ανώτατα δικαστήρια θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα συνταγματικά. Ένα άλλο θέμα που αναφέρεται στην έκθεση έχει να κάνει με τη συμμετοχή του Εθνικού Μεσαισιωτικού Δικαστή ε, σε επίπεδο ένωσης ε, στις ε, διάφορους, διάφορους σχηματισμούς, στις διάφορες συνθέσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και ουσιαστικά πρέπει να συμμετέχει ο δικαστής που έχει διοριστεί δυνάμει αυτού του κράτους στις, ε, στην εξέταση των υποθέσεων έναντι κάποιου ε, θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συμμετέχει ένας εκλεγμένος δικαστής ε, ε, εκπροσωπώντας ε, την Ένωση. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με τις ιδιωτηρότητες του δικαίου της Ένωσης ε, που θίγουν τη συγκεκριμένη υπόθεση και φυσικά δεν πρέπει να είναι ένας ad hoc δικαστής αλλά ένας μόνιμος δικαστής ο οποίος θα είναι πλήρως απασχολούμενος και φυσικά αυτό με το σκοπό να γνωρίζει πολύ καλά και από την εκ των έσω του δικαστηρίου πώς επιλύονται οι διάφορες προσφυγές κατά των κρατών και να έχει στη διάθεσή του και τα απαραίτητα στοιχεία σύγκριση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιδέα περιλαμβάνεται στο σχέδιο ψηφίσματο που έχουμε ενωπεί. Όμω, όταν αναφέρεται ότι ο δικαστή που εκλέγεται ε, εξ ονόματο τη Ένωση θα πρέπει να είναι ισότιμο με του υπόλοιπου δικαστέ. Είναι επίση προφανέ ότι η Ένωση θα έχει δικαίωμα να παρουσιάσει με ένα κατάλογο ίδιων υποψηφίων για την εκλογή ενό εξ αυτών ω δικαστή εξ ονόματο τη Ένωση. Αν συνεχίσουμε τώρα με την εξέταση των περιπτώσεων κατά τις οποίες θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εναγόμενη σε διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι οριστικές αποφάσεις, οι τελεσίδικες αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου θα πρέπει να έρχονται σε γνώση του Συμβουλίου Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ώστε να προχωρούν στην εκτέλεσή τους. Όπως γνωρίζετε αυτή η Επιτροπή είναι το ανώτατο διακυβερνητικό όργανο το οποίο απαρτίζεται από τους πρεσβευτές των κρατών μελών ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίοι υποκαθιστούν, αντικαθιστούν τους υπουργούς τους. Όταν πρόκειται βέβαια για την εφαρμογή μιας απόφασης η οποία διαπιστώνει μια παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων από ένα φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ψήφου από την πλευρά του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρεται εκπεφρασμένα στο σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε ενωπιών μας. Και τονίζω ιδιαίτερα το ότι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχει, να συμμετέχει επίσης και στη συνεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου εξετάζεται η, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων εναντίον δεδομένων κρατών μελών. Αυτό, επομένως, είναι ορθό, διότι με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα να δίδεται στον εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης το σύνολο των επιχειρημάτων και αιτιολογήσεων αυτής της απόφασης. Τώρα, σε σχέση με το θέμα του σε ποια νομικά εργαλεία θα πρέπει να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της ε, σύμβασης, και εδώ φυσικά περιλαμβάνει και τα πρωτόκολλα 11 ή 14 ή ακόμα πρέπει να συμμετέχει σε πρωτόκολλα τα οποία είναι για τα οποία είναι προαιρετική η προσχώρησή της. Ξεκινώντας από την ιδέα ότι καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υποχρεωμένη να προσυπογράψει αυτά τα νομικά εργαλεία, τα οποία είναι προαιρετικού χαρακτήρα, θεωρώ ότι είναι σωστή η πρόταση που γίνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιοριστεί μονάχα στα πρωτόκολλα 1, 4, 7 και 12, τα οποία περιλαμβάνουν σημαντικά δικαιώματα. Κάποια από αυτά είναι δικαιώματα τα οποία μπορούν πράγματι να παραβιαστούν με συγκεκριμένο τρόπο από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συγκεκριμένα δικαιώματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διακρίνει το ιδιαίτερο συμφέρον των πολιτών της. Επίσης θα πρέπει να δούμε αν αυτή η προσχώρηση θα γίνει μέσω μιας ανεξάρτητης συμφωνίας ή αν θα είναι ένα νέο πρωτόκολλο που θα τροποποιεί τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τι Θεμελιώδει Ελευθερίε. Και οι δύο δυνατότητε είναι ανοιχτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να καθυστερήσει αυτή η προσχώρηση μετά από την 1η Ιουνίου 2010 που είναι η ημερομηνία στην οποία θα τεθεί σε εφαρμογή το πρωτόκολλο 14 και η τροποποιημένη αντιστοίχω μορφή τη σύμβαση. Η λογική μια τέτοια αντιμετώπιση είναι ότι αυτό το κείμενο το οποίο θα είναι τροποποιημένο προβλέπει και τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ούτω ή άλλως ότι θα είναι χρήσιμο να αποφύγουμε στο βαθμό του δυνατού το να υπάρχει πολυπικιλία και πολυμορφία και πολλαπλότητα εργαλείων νομικών γιατί θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να ενσωματώσουμε με παγιοποιημένο τρόπο τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες. Μετά από όλες αυτές τις προηγούμενες σκέψεις τις οποίες σας έχω παρουσιάσει, που είναι επιλεκτικές και γενικές, θα ήθελα να σταθώ τώρα σε ένα τμήμα του ψηφίσματος, το οποίο κατά την άποψή μου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και για την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας δικαίου, της ενισχυμένης ασφάλειας δικαίου, που θα πρέπει να πριτανεύει μετά από την προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Ρώμης. Πρόκειται για, το 11, για την ενδέκατη παράγραφο όπου υπάρχει μνήα στα προβλήματα με τα οποία αντιμετωπίζει το σύστημα της σύμβασης της ε, Ρώμης και που αναφέρεται επίσης στην ανάγκη να υπάρξει μια κατεπίγουσα μεταρρύθμιση αυτού του συστήματος λόγω της ε, πλημμυρίδος ουσιαστικά προσφυγών που έρχονται στο δικαστήριο. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2009 ο αριθμός αυτών των προσφυγών ήταν 119.298 οι εκρεμείς προσφυγές για κάποιο σχηματισμό αυτού του δικαστηρίου. Είναι γεγονός ότι το πρωτόκολλο 14, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στην 1η Ιουνίου του 2010, είχε σαν στόχο να βελτιώσει την παραγωγικότητα του δικαστηρίου, αλλά εξάλλου αληθεύει επίσης <clears throat> ότι αυτή η βελτίωση δεν απεδείχθη επαρκής. Μόνο 20 με 25% θα, τα 100 θα αυξήσει την παραγωγικότητα του δικαστηρίου κατά την άποψη του ίδιου του δικαστηρίου όπως περιγράφεται στην ετήσια έκθεσή του του 2009. Το πρωτόκολλο 14 ουσιαστικά κατανέμει τις προσφυγές μεταξύ του ίδιου αριθμού δικαστών με την πρόβλεψη ότι σε ορισμένου σχηματισμού του δικαστηρίου θα μπορέσουν να μειωθούν οι προσφύγες, αλλά χωρί κάποια εγγύηση για κάτι τέτοιο. Με τον τρόπο αυτό είναι περιορισμένη η εφαρμογή του άρθρου 14, του πρωτοκόλλου 14. Τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη έχουν λάβει γνώση αυτού του θέματο, και γνωρίζουμε ότι στις 18-19 του Φεβρουαρίου έγινε στο Ιντερλάκεν μια διυπουργική σύνοδος για να αντιμετωπιστεί το μέλλον του συστήματος προσφυγών προέκυψε ένα ενδιαφέρον σχέδιο δράσης από αυτή τη συνεδρίαση που ελπίσουμε ότι θα αποδώσει τους προσδοκούμενους καρπούς. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε υπερβολικές και φρούδες ελπίδες. Αυτοί οι καρποί δεν μπορούν να επιτευχθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, σας υπενθυμίζω ότι προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα της μεταρρύθμισης και εις βάθος του συστήματος του Ευρωπαϊκού Καστηρίου επέτρεψα στον εαυτό μου και να μακρηγορήσει ακόμα γιατί αυτή η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει την νομική ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα θέματα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως απαιτεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Ραμόν Χαουρεγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει την απαραίτητη επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είναι απαραίτητο να συμμετάσχει στην μεταρρύθμιση και στην βελτίωση των συνδικών στο Δικαστήριο του Στασβούργου. Σας ευχαριστούμε καθηγητά για την έκθεσή διαβάσετε από ό,τι είδα και ένα κομμάτι τη ομιλία. Αν υπάρχει κείμενο γραπτό, θα μπορούσε να μοιραστεί ή να μπορούσε να μπει στα πρακτικά. Εν πάση περιπτώσει, όσο σύντομη και να είστε υποχρεωμένοι να είναι, αφήστε μα τα γραπτά κείμενα, αν τα έχετε, γιατί είναι σημαντικό για μα. Για να τηρούμε το χρόνο των 15 λεπτών μιλητή, στα 14ο λεπτό θα χτυπάω δύο, δύο χτυπήματα με το σφυράκι μου για να ξέρετε ότι πλησιάζει το πέρας της ομιλίας σας. Ο καθηγητής Αντώνιο Παπίσκα, καθηγητής του Πανεπιστήμα της Πάντεβα. Στην έδρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και η ειρήνη έδρα της UNESCO. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Έχουν γραφτεί πολλά για το θέμα αυτό και εγώ θα συνοψίσω μερικές ιδέες. Πολύ σύντομα θα σας παρουσιάζω μια συστημική περιγραφή του συστήματος. Μια κατράμε τη σημασία του εγχειρήματο. Μετά θα πω μερικά θέματα για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Με την προσχώρηση στη συνθήκη η Ένωση τυπικά εισάγεται μέσα στα πιο προθυμένα περιφερειακά συστήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βέβαια, ήδη ε, έχει αρχίσει να μπαίνει στο παγκόσμιο σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν υπέγραψε την σύμβαση της UNESCO για την προστασία της ε, πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων και μετά όταν διαπραγματεύθηκε την προσχώρηση στην σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε ένα άνοιγμα δηλαδή της Ένωση σε θέματα διεθνούς δικαίου, γενικού δικαίου αφορά τους ανθρώπους. Αλλά η συμμετοχή της Ένωσης στα δύο αυτά συστήματα, περιφερειακό της Ευρώπης και παγκόσμιο, θα ενισχύσει φυσικά και το ένα και το άλλο. η προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση είναι ένα ιστορικό γεγονός που ξεπερνάει την Ευρώπη. Γιατί το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα κερδίσει και σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ και μερικά χρόνια στα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργάνων Υπάρχει η αναφορά σε αυτό που λένε International Rule of Law, διεθνής κανόνας δικαίου, που πρέπει να ισχύει στις διεθνείς οργανώσεις, όχι μόνο για τα κράτη. Ε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υλοποιήσει πλήρως αυτή την αρχή υποκείμενη στην, στην δικαιοδοσία ενός υπερεθνικού δικαστηρίου που είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επομένως, η προσχώρηση δεν είναι μόνο θέμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ δύο μεγάλων παγκοσμίων θεσμών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προσχώρηση Ένωσης που είναι μια ενότητα sui generis με υπερεθνικά δικαιώματα σημαίνει ότι θα υπόκειται σε μια άλλη υπερεθνική αρχή, δικαστήριο του Στρασβούρου, που γίνεται υπερ-υπερεθνική στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Αυτά για την εγγύηση της πολύπλοκης αυτής δομής. Φυσικά το κείμενο της ομιλίας μου θα σας το δώσω μετά. Συνοψίζω αρκετά γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο ραντεβού των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο της Ευρώπης με ένα κεκτημένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό το κεκτημένο. Αναφέρομαι στο κείμενό όμως αυτό με λεπτομέρειες. Ας θυμηθούμε όμως το πώς ξεκίνησε αυτό το κεκτημένο. Το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος του Αλτιέρο Σπινέλη. αν πάρετε το άρθρο 4 αυτού του σχεδίου συντάγματος θα βρείτε σε μια πρώτη μορφή αυτό που βλέπουμε τώρα στις ε, ε, μετέπειτα συνθήκες και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν πάση σε αυτό το κεκτημένο της Ένωσης υπάρχουν τα άρθρα τίτλος 1 και 2 των τροποποιητικών συνθήκων όπου αναφέρεται ότι η Ένωση στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δική μου η ερμηνεία είναι ότι το άρθρο 2 της τροποποιητικής συνθήκης είναι ο γενικός κανόνας, ο οποίος συνοψίζει στη συνταγματική της διάσταση τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης, που με τη σειρά τους όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα προωθούν σε ανώτερο επίπεδο νομικής δέσμευσης την χάρτα των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην χάρτα του 89. Εδώ υπάρχει ο, ο γενικός κανόνας των πρωτογενών κανόνων της Ένωσης. Τώρα, η διομορφία η πολιτιστική ιδιομορφία της Ένωσης η προστασία δηλαδή της ταυτότητας της Ένωσης και της νομικής ιεράρχησης σε θέματα Ένωσης. Εδώ ενδιαφέρον έχει το πρωτόκολλο 8 όπου θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται η ανάγκη προστασίας των δικών χαρακτηριστικών της Ένωσης και των δικαιωμάτων της Ένωσης. Κάνουμε διάκριση δηλαδή ανάμεσα στην ταυτότητα της Ένωσης στο σύνολό της και της νομικής τάξης της Ένωσης. Η ταυτότητα της Ένωσης είναι το πολιτιστικό, θρησκευτικό και ανθρωπιστικό στοιχείο κληρονομιά της Ένωσης από την οποία προέρχονται οι καθολικές αξίες που αποτελούν τα απαραβίαστα δικαιώματα του προσώπου, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, όπως τα ορίζει το προήμιο της ε, μεταρρυθμιστικής συνθήκε. Επίσης, η πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά της Ένωσης αναφέρεται και ανάπτυξη κοινών αξιών με σεβασμό της πολυμορφίας, πολιτισμού κλπ. Η φράση «unity in the diversity» στα αγγλικά, η πολυμορφία στις αξίες, ουμανιστικού χαρακτήρα που στηρίζει την αξιοπρέπεια του ατόμου και στο σεβασμό της ακυριότητας του ατόμου και ως πνευματικού όντως της οικογένειας, τη θέση του στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η προστασία λοιπόν αυτής της δημορφίας, πολιτιστικής δημορφίας της Ένωσης πέρα από το νομικό κείμενο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο παραρτήματος με μορφή διακήρυξης όπου θα αναφέρεται το ότι η Ένωση από το 2007 αποτελεί προσχώρηση στις συνθήκες της πολιτιστικής της προστασίας δύο πρακτικές προτάσεις. Πρακτικές υποδείξεις, λοιπόν, διαδικασία για την προσχώρηση ορίζεται σαφώς στο άρθρο 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης, Κομισιόν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Το εργαλείο προσχώρησης, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να, είναι, να έχει μορφή συνθήκες και όχι πρωτοκόλλου, για λόγους τυπικούς γιατί είναι νομική προσωπικότητα η Ένωση στο ύψος κρατών. Στο προήμιο της συνθήκης προσχώρησης θα πρέπει να αναφέρεται η πρωτογενή σπηγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν τα βλέπουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 50 γιατί είναι το μόνο περιφερειακό σύστημα στην Ιδρυτική Σύμβαση που δεν αναφέρεται ρετά στις πρωτογενείς πηγές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ αυτή την αναφορά τη βρίσκουμε στη Σύμβαση των, στις Αμερικής, Αφρικής, Αράβων κλπ. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να τονίσουμε την ορθοδοξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σωρίζονται ως πρωτογενής νομική πηγή. Η προσχώρηση στο πρωτόκολλο της συνθήκης δεν θα έπρεπε να είναι αυτόματη. Θα πρέπει να γίνεται διάκριση ανάμεσα στα πρωτόκολλα που αναφέρονται σε προστατευόμενα δικαιώματα από τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τα πρωτόκολλα που έχουν επικυρωθεί από όλα τα κρατημέλη και τα πρωτόκολλα που έχουν εν μέρη επικυρωθεί. Δίκαστης της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενδεχομένως. Θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και δύο ή τρεις, θεωρώντας ότι με την προσχώρηση στη συνθήκη, στη σύμβαση, ε, θα αυξηθεί πάρα πολύ το έργο του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Ο δικαστής της Ένωσης θα πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τις ιδιομορφίες, τις πολιτιστικές φυσικά, που είναι πολιτικά, αστικά, πολιτιστικά και άλλα δικαιώματα στην Ένωση. Η Ένωση να μπορεί να προσφύγει ως διάδικο στο δικαστήριο του Στρασβούργου, να μπορεί να συμμετέχει παράγγελα με το κράτος μέλος, κατά κύρια αρχή και αντιστρόφως συμμετοχή στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην Επιτροπή Υπουργών η εκπροσώπηση της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του πολίτη στην κοινοβουλευτική συνέλευση να εκπροσωπείται από μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τελειώνω. Θεσμοί και διαδικασίε μη, μη ε, δικαστηριακού χαρακτήρα, ombudsman, ε, διαμεσολαβητέ, εθνικέ επιτροπέ κλπ. σε μια διακήρυξη, ένα πρωτόκολλο, παράτημα, στη, στη σύμβαση προσχώρηση, στη συνθήκη προσχώρηση, θα πρέπει να υπάρχουν αυτά ω εγγύηση και για να ελευθερωθεί το έργο του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και το έργο του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπίσκη, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε διπλά και για το πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο της παρουσίασής σας και γιατί μας κάνατε να κερδίσουμε και πέντε λεπτά σε σχέση με το χρόνο που είχε καθοριστεί εξ αρχής. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να διακόψουμε την ακρόαση των πυρογνωμόνων και να περάσουμε στη συζήτηση, να ακούσουμε τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Έχουμε στη διάθεσή μας 15 λεπτά. Βλέπω ότι ο κύριος Τερβίγκο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, καθηγητές ε, Παστόρ, Ριδρουέχο και Παπίσκα. Πραγματικά ε, ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικές οι παρεμβάσεις τους γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι αυτοί τα πράγματα και μπορούν να μας βοηθήσουν για να δούμε πως και εμείς μπορούμε να συνδράμουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τα πολύπλοκα θέματα αυτής της προσχώρησης. Γιατί εμείς σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσαμε μάχη για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση εδώ και πολλά χρόνια το ανέφερε και ο κύριος Παπίσκα από το έγγραφο Σπινέλη. Τότε υπήρχε η φιλοδοξία αυτού του Κοινοβουλίου για την προσχώρηση και πάντοτε εμείς σκεφτόμασταν ότι η προσχώρηση θα ήταν το τέλος του ταξιδιού. Αναφέρθηκε από τον κύριο Παστόρ ε, η ζωτική κατάσταση, η κριτική κατάσταση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτή η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Σύμβαση είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κριτική κατάσταση. Με ποιο τρόπο η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορεί να σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε στην επίλυση προβλημάτων. Ποια πρέπει να είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα αυτά θα ήθελα να εμβαθύνετε κάπως περισσότερο και το αναφέρετε γιατί εγώ από τη δεκαετία του 80 που ασχολιόμουν με θέματα του Συμβουλίου της Ευρώπης νομίζω ότι τα έχω ξεχάσει κάπως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η αγκαιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι τίθενται πολύ συγκεκριμένα ζητήματα όταν ε, εμείς νομοθετούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τα μεταφέρουμε όλα στην εθνική νομοθεσία και όλες ε, ε, οι αποφάσεις, κυρίως οι εθνικές αποφάσεις και όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε σκεφτούμε ίσως τις περιπτώσεις για τις οποίες οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι αντικείμενο αυτού του δικαίου. Γιατί, ξέρετε, έχουμε μία σειρά περιπτώσεων όπου έχουμε τα κράτη-μέλη που έχουν θέσει σε εφαρμογή αυτές τις οδηγίες και πρέπει να αναρωτηθούμε αν είναι τα υποκείμενα στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, θα ήθελα να μου πείτε ε, η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι ακριβώς σημαίνει. Ο κύριος Χαράγουι. Από, αν ε, κατάλαβα καλά, πώς είπε ο κύριος ε, Παπίσκα, εσείς είστε υπέρ του να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει δηλαδή. Εμείς, ε, εμείς θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη είναι παρόντα Η Μία πρόσθετη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τέτοια στην κοινοβουλευτική συνέλευση δεν θεωρούμε απαραίτητη. Και είναι αλήθεια ότι τίθεται το πρόβλημα ότι στην εκλογή των δικαστών θέλουμε να <laughs> παρευρισκόμαστε, αλλά δεν είδαμε πώ μπορούμε να το συνδυάσουμε αυτό με συγκεκριμένη παρουσία στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Μπορείτε να μου το ξεκαθαρίσετε αυτό το θέμα. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο μέχρι τώρα. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική άσκηση στην οποία αποδιόμαστε σήμερα. Θα πρέπει όμως να θυμούμαστε <clears throat> ότι η απόφαση για να προσχωρήσουμε, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να προσχωρήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες, είναι το αντιστάθμισμα ή πίν για την απόφαση να δεχτούμε να γίνει δεσμευτική χάρτα ανθρωπινών δικαιωμάτων ω τμήμα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Κάποιοι από εμά που ήμασταν παρόντες στην συνέλευση η οποία συνέταξε τη χάρτα αυτή και την νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θυμόμαστε πόσο ευαίσθητο ήταν το θέμα αυτό για πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και το κράτος μέλος από το οποίο εγώ προέρχομαι και έχω την καλύτερη γνώση αυτού για τα θέματα αυτά και που έχει αντισταθεί σε μεγάλο βαθμό στον υποχρεωτικό χαρακτήρα της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κατά παράδοξο τρόπο, λέει η συνθήκη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει μέλος <clears throat> στη σύμβαση αυτή, λες και είναι κάτι τότε τελεσμένο. Αλλά επίσης και ανοήτως φοβάμαι ότι πρέπει να πω, ήταν αυτό μια παραχώρηση η οποία έγινε μετά από το γαλλικό και ολλανδικό δημοψήφισμα που δεν δέχτηκαν την μορφή που είχε συνθήκη το 2004. Στη συνέχεια λέγεται με παράλογο όπως είπα τρόπο ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί με ομοφωνία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και φυσικά και με την ε, σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι στα πλαίσια της περαιτέρω διερεύνησης αυτού του θέματος θα εξασφαλίσουμε και μια ισχυρή συνένεση μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο για να προωθηθεί το θέμα αυτό και θα ήθελα να ακούσω και από τους ειδικού μας εδώ κατά πόσον πιστεύουν ότι μπορούν να ανακύψουν θέματα διαφωνιών μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία θα μπορούσαν να περιπλέξουν τη λήψη μιας απόφασης για να προσχωρήσουμε πράγματι στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά δεύτερο λόγο, <clears throat> θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω από τους εμπειρογνώμονες ποια είναι η κρίση τους σε σχέση με το αν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η ποιότητα και το σθένος αυτής της χάρτας μπορούν να τύχουν πλήρους προστασίας αν εμεί προσχωρήσουμε στη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και κατά τρίτο λόγο, σε σχέση με την Υπουργική Σύνοδο, την Επιτροπή Υπουργών. Συμφωνούμε εδώ ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να είναι το όργανο το οποίο θα έπρεπε να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα θέμα όπου πρέπει και το Κοινοβούλιο να κάνει ακουστή τη γνώμη του και να τα διελευκάνει αυτά τα θέματα. Να προσθέσω κι εγώ μια ερώτηση. Ο, ουσιαστικά έχει να κάνει με τις δύο παρεμβάσεις που ακούσαμε και φαντάζομαι ότι και πολλοί εμπειρογνώμονε ε, μπορούν να παρεμβούν, όχι μόνο τα μέλη του Κοινοβουλίου. Στο άρθρο 6 της Συνθήκης Λισαβόνας λέγεται ότι η προσχώρηση δεν τροποποιεί τις αρμοδιότητες ε, της ε, Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ποια όρια τίθεται. Πρόκειται για ένα κανόνα που δεν διαφέρει σε σχέση με αυτή που έχουμε στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο δεύτερο εδάφιο λέει ότι οι διατάξεις ε, της ε, χάρτας δεν επεκτείνουν σε καμία περίπτωση ε, την δικαιώματα της Ένωσης. Όμως υπάρχει ένα όριο τώρα στην εφαρμογή της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή όχι. Ποιος θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σταθώ στο ερώτημα το οποίο ετέθη από τον Ινίγκο Μέντες Δεβίγο σε σχέση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, η λέξη σε κρίσιμη κατάσταση, σε δύσκολη κατάσταση αναφέρεται ήδη στην έκθεση, στην αιτήσια του δικαστήριου αν θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει πλήρως στη σύμβαση. Εγώ νομίζω ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης η οποία είναι απαραίτητη για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια μεταρρύθμιση σε βάθος, σε τελική ανάλυση εξαρτάται από την πολιτική θέληση των εμπλεκομένων μερών. Υπάρχουν προφανώς τεχνικά προβλήματα, αλλά αυτά μπορούν να επιληθούν μονάχα εάν υπάρξει η απαραίτητη πολιτική θέληση όλων των εμπλεκομένων. Πιστεύω λοιπόν ότι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πολιτική θέληση για τη μεταρρύθμιση. Και επομένως από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει την επίλυση των προβλημάτων του ΕΔΑΔ. Μπορεί να μην ισχύει αυτό για όλα τα κρατημέλη εξίσου στο Συμβουλίο της Ευρώπης και μπορώ να αναφέρω την περίπτωση της Ρωσίας. Δεν είναι πρόβλημα να κατονομάσω μια χώρα η οποία έχει καθυστερήσει την εφαρμογή του πρωτοκόλου 14. Δυστυχώς νομίζω ότι μια τέτοια αντιμετώπιση μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον όταν πρόκειται για τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου του ΕΔΑΔ. Φοβάμαι ότι θα είναι απαραίτητο να υπάρξει και πολιτική θέληση από άλλες χώρες, αλλά σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αμελήσει να έχει την απαραίτητη πολιτική θέληση. Ετέθηκε ένα άλλο ερώτημα από κάποιον ομιλητή για το κατά πόσο η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση είναι απαραίτητη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουν θέσει πάρα πολλοί. Πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλές προσωπικότητες. Αυστηρά ενία δεν είναι απαραίτητο, γιατί ήδη εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που είναι μέσα στο δεσμευτικό της εσωτερικό δίκαιο και εφόσον εφαρμόζεται αυτή η χάρτα από τα Εθνικά Δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά το σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν ενισχυθεί όμως αυτό το πλαίσιο με την προσχώρηση τη Σύμβαση της Ρώμη και την αποδοχή της δοσιδικίας του ΕΔΑΔ, αυτή η νομική ασφάλεια, η ενισχυμένη όπω είπα νομική ασφάλεια, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για αυτό το βήμα. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία να ενισχύσουμε ακόμα αυτή την ασφάλεια δικαίου η οποία υπάρχει φυσικά μετά την συνδίκη της Λισαβόνας και μπορούμε όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι σαν Ευρωπαίοι πολίτες με αυτή την προοπτική. Αυτά ήθελα να αναφέρω σε σχέση με τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Για την προσχώρηση, ναι, η προσχώρηση λέμε ότι είναι απαραίτητη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθεαυτή είναι ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει εγγυήσει στο εσωτερικό της. Αλλά επιπλέον θα υπάρχουν και εγγυήσει οι πρόσθετες που παρέχονται από ένα υπερεθνικό σύστημα, όπως είναι το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό το να υπάρχουν αυτές οι πρόσθετες προσχώρηση στη σύμβαση ενισχύει τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και φυσικά δημιουργεί τους πολίτες. Μιλάμε εδώ για μια τελειοποίηση αυτής της διαδικασίας βελτίωσης ε, των ε, νομικών και πολιτικών συστημάτων. Το άρθρο 6 της συνθήκης τώρα. Δεν τροποποιούμε τις αρμοδιότητες της Ένωση, Εν τω μεταξύ, οι αρμοδιότητες της Ένωση εμπλουτίζονται στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λόγω χάρη προστίθενται και τα κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιώματα. Ο κοινωνικό χάρτη έχει πλήρη νομική αξία. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση στι αρμοδιότητε του Δικαστηρίου τη Ένωση εκεί ε, συμπεριλαμβάνονται και τα κοινωνικά δικαιώματα. Είναι αρμοδιότητά του, δεν είναι αρμοδιότητα του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να τη διατηρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμμετοχή στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαφορετική κατάσταση έχουμε εκεί με την περίπτωση του δικαστή. Εκεί, στο δικαστήριο της Ένωσης, εκεί είναι πλένο γιούρα. Εδώ έχουμε συμμετοχή ad hoc, γιατί η εκλογή του δικαστή έχει άλλο βάρος, ε, αν θέλετε, στην ουσία πέρα από την εκπροσώπηση ad hoc. Εγώ βλέπω το θέμα του εκδημοκρατισμού των διεθνών θεσμών, του συστήματος διεθνών σχέσεων. Έτσι λοιπόν ε, εδώ ενισχύουμε την διεθνή δημοκρατία. Ποιο είναι το βάρος ε, τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσχωρεί στη σύμβαση ε, στα πλαίσια των εργασιών του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Εδώ θα πρέπει να προβλέψουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδράμει το Συμβούλιο της Ευρώπης με ανθρώπινους πόρους και υλικούς πόρους. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό στο πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και περνάμε στο δεύτερο γύρο της ακρόασης μέχρι τις 11 η ώρα με παρεμβάσεις του καθηγητή Νόμπελ Πολ Έγγελ εκδότη του Ευρωπαϊκού Εφημερίδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του καθηγητή Ζαν Πολ Ζακ από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και διευθυντή στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και τον καθηγητή Όλιβερ Ντεσίτε, καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Νεύ. Αρχίζουμε με τον καθηγητή Νόρμπερτ Πολ Έγγελ. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Θέλω να τονίσω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ μεταξύ όλων αυτών των εμπειρογνωμόνων και των ομομαθών και να παρουσιάσω την απόψή μου. Εγώ δεν είμαι καθηγητής, έχω ένα επίτιμο διδακτορικό απλώς και ουσιαστικά εγώ είμαι εκδότης μιας εφημερίδος που ασχολείται με πολιτικά και νομικά θέματα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εδώ είναι το θέμα της διοικητικής ανεξαρτησίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να προκύψουν με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν μιλάμε τώρα για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά σε ένα οικοδόμημα συμβατικό, όπου θα σημαίνει αυτό ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα αντιμετωπίζονται με ένα ιεραρχικό τρόπο, αλλά ότι τα μέλη τα οποία έχουν προσυπογράψει τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όλα από κοινού θα εξετάζουν την προστασία και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη που έχουν προσυπογράψει αυτή τη σύμβαση. Επομένως, εδώ δεν είναι πια ένα θέμα κρατικής υπόστασης και ιεράρχησης. Για μένα, τα πλεονεκτήματα μπορούν να συνοψιστούν σε τρία σημεία. Πρώτον, βελτίωση της ε, πολιτικής νομιμότητας και νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 250 αναφέρεται στην ε, χάρτα ανθρωπινών δικαιωμάτων. Δηλαδή η αιτιολόγηση και ο Ζαν Πολ Ζακέ μπορεί να με διορθώσει αν δεν τα λέω σωστά. Στην αιτιολόγηση λοιπόν του προημίου αναφέρεται όχι μόνο το θέμα αυτό, αλλά, της ε, χάρτας, αλλά και η νομολογία και η εφαρμογή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Επομένω, η η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, βάσει της ε, χάρτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρήματων, βασίζεται στην ομολογία και την εφαρμογή του ΕΔΑΔ. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έστω και έμεσα μέσω των κρατών μελών, μέσω των κρατών μελών που έχουν προσυπογράψει τη Σύμβαση για τα Ανθρωπίνα Δικαιώματα, δεσμεύεται από τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Αναφέρομαι στην απόφαση Βόσφορος, η οποία παίζει κάποιο ρόλο σε, στις σημερινές συζητήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει την ομολογία η οποία έχει παραχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και η οποία φτάνει σε ένα σημαντικό επίπεδο ποιότητας. Λέει ότι υπάρχει η παράλληλη αξία και ισοτιμία των αποφάσεων του Λουξεμβούργου, του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, αλλά λέει ότι είναι ανασκευάσιμη κατά κάποιο τρόπο η νομολογία του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου και να ζητήσει επανεξέταση μιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα μέσω αυτή τη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Ένωση από ένα απλώ αντικείμενο δικαίου να γίνει ένας σημαντικός παίκτη στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έρχομαι τώρα πάλι και στο θέμα τη ανεξαρτησίας του ΕΔΑΔ. Μιλάω για την διοικητική ε, ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τη στελέχωση και επίσης σε ό,τι αφορά την αυτονομία σε επίπεδο προπολογισμού. Αυτό το οποίο βλέπω σε αυτή την πρόταση, στο ψήφισμά σας, είναι η προϋπόθεση που θέτεται, που πρέπει να είναι επαληθεύσιμη, πρέπει να είναι εκπληρώσιμη, πρέπει δηλαδή να, γίνεται, να μπορεί να γίνει αυτή η προσχώρηση σε ένα βραχή χρονικό διάστημα και χωρίς οικονομικό κόστος. Επομένως, με βάση αυτή την προϋπόθεση δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ώστε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα προβλήματα τα οποία είναι διοικητικού χαρακτήρα. Και εκπλήσωμαι εδώ όταν βλέπω ότι ο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, και μιλάω τώρα σε θεσμικό επίπεδο, από τότε που υπάρχει το μόνιμο αυτό δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το 1989 δηλαδή, αντιμετωπίζει το θέμα της, του προσωπικού και της τελέχωσης σαν ένα θέμα εξουσίας. εγώ χάρη στην καγκελαρία του δικαστηρίου, έχει μείνει, την έχει αφήσει κενή επί ένα χρόνο, διότι ο Γενικός Γραμματέας ήθελε να υποχρεώσει το ΕΔΑΔ να ακολουθήσει τη δική του πολιτική προσωπικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπετε και, στο, και στα πρακτικά της κοινοβουλευτικής συνέλευσης, όπου ο τωρινός Υπουργός Δικαιοσύνης τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανίας και άλλοι βουλευτές είχαν θέσει ερωτήματα σε σχέση με αυτή τη συμπεριφορά και κατά την άποψή μου δεν πήραν μια, μια επαρκή απάντηση από το Γενικό Γραμματέα της κοινοβουλευτική Συνέλευσης. Δεν πρόκειται για το ότι ένας δικαστής δεν μπορεί να έχει έλεγχο του προσωπικού του, ήδη είναι ένα πρόβλημα. Αλλά το να αποφασίσει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ποιος θα είναι ο συνεργάτης του, αυτό είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τα εσκαμένα. Νομίζω ότι για να υπάρξει αποτελεσματική λειτουργία του δικαστηρίου χρειάζεται το κατάλληλο περιβάλλον σε διοικητικό επίπεδο. Και δεν μπορεί κανείς να έχει στην πλάτη του μια ανοιχτή πόρτα, για να το πω έτσι, όταν εργάζεται σε ένα γραφείο. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι σημαντικά τα διοικητικά θέματα. Αν δείτε το θέμα επίσης και από πολιτική έποψη ο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου τη Ευρώπη επιλέγεται σε πολιτικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Το ξέρουν αυτό όλοι οι βουλευτέ βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει κανεί να εκλεγεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να παρουσιάσει τον εαυτό του, θα πρέπει να κάνει τα απαραίτητα διαβήματα, θα πρέπει να δεσμευτεί να πράξει το Α ή το Β, να αναλάβει δεσμεύσει εναντίον ομάδων, είτε είναι κοινοβουλευτικέ ομάδε είτε είναι εθνικέ ομάδε κτλ. Και ένα άτομο το οποίο επιλέγεται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ένα άτομο το οποίο αναγκάζεται να παίξει αυτό το ρόλο μιας εξισορρόπησης, αν θέλετε, πολιτικών τάσεων μέσα στο, στο δικαστήριο, το να πάρει αυτό το άτομο την ικανότητα να ασκεί μια πολιτική προσωπικού σε ένα δικαστήριο αυτό σε διεθνές επίπεδο είναι κάτι το αρκετά ασυνήθιστο. Στην περίπτωση του, του, γερμανικού, όμως, του συνταγματικού δικαστηρίου υπήρξε αντίδραση στο να υπάρχει μια τέτοια παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αντίστοιχα έχει ακολουθηθεί η ίδια πρακτική και στην περίπτωση του Αυστριακού Ανώτατου Δικαστηρίου να λαμβάνονται λοιπόν αποφάσεις και να επιβάλλονται από άλλους φορείς σε σχέση με τη στελέχωση σε προσωπικό. Για μένα λοιπόν μια σημαντική προϋπόθεση για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι το ΕΔΑΔ θα πρέπει να εξασφαλίσει την συνήθη ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά το προσωπικό του. Αυτό δεν είναι ένα προπατορικό σφάλμα του δικαστηρίου. Δεν ξεκίνησε έτσι το ΕΔΑΔ. Είναι όμως κάτι το οποίο προέκυψε στο δρόμο της λειτουργίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επομένως, πρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργήσε η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στην αρχή υπήρξε η εκπόνηση αυτής της σύμβασης στη δεκαετία του 1950, με στόχο να υπάρχει και μια δυνατότητα δικαστικής προσφυγής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα κράτη-μέλη δεν προχώρησαν τόσο πολύ ώστε να φτάσουν να πούν ότι έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δικαστήριο. Όχι, είπαν ότι με μια Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ατομικέ προσφυγέ και η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τα νομικά ερωτήματα, να κάνει εξέταση των πραγματικών στοιχείων. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να γίνουν και να καλύψουν αυτά τα θέματα, αυτά πάντα και κλεισμένα των θυρών, χωρίς να υπάρχει παρουσία του κοινού και επί τη βάση των εκθέσεων οι οποίες θα παραγόντουσαν και θα εξεταζόντουσαν στην Επιτροπή των Υπουργών θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε ή όχι μια ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ το δικαστήριο το οποίο συγκροτήθηκε μόνο αργότερα μετά από την πρώτη λειτουργία της Επιτροπής των Υπουργών στην αρχή έπαιζε μονάχα ένα επικουρικό ρόλο. Μπορούσε να γίνει η επίκληση του δικαστηρίου μονάχα όταν το ζητούσε ένα κράτος μέλος ή όταν η Επιτροπή των Υπουργών ζητούσε να υπάρξει προσφύγει στο δικαστήριο. Επομένω, στην αρχή είχε πολύ περισσότερο προσωπικό η Υπουργική Επιτροπή από ότι το ίδιο το δικαστήριο. Και στο παλιό κείμενο ε, της σύμβασης, το άρθρο 37, έλεγε ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι αυτός ο οποίος επιλέγει τους συνεργάτες της Επιτροπής. Ανέφερε ότι η γραμματεία εξασφαλίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επομένως αυτός είχε το δικαίωμα να επιλέγει το προσωπικό το οποίο θα στελέχωνε αυτήν την Επιτροπή. Για την ε, στελέχωση του δικαστηρίου δεν ισχύει τίποτα τέτοιο και δεν έχει το χαρακτήρα του ανώτατου διοικητικού αξιωματούχου του δικαστηρίου ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι σαφές λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στα πλαίσια της αυροφροσύνης θα έπρεπε να κάνει σαφές προς το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι η έγκριση της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα εξαρτιόταν από την εξασφάλιση της παραδοσιακής σε παγκόσμιο επίπεδο ανεξαρτησίας του δικαστηρίου και του προσωπικού του. Στην περίπτωση του, αμερικανικού, του διαμερικανικού μάλλον δικαστηρίου στην Κωνσταντίνα για υποθέσεις μεταξύ Αμερικανικών κρατών, ετέθη πράγματι αυτό το θέμα. Και όπου με μία γραπτή ε, διαθεσμική συμφωνία επελήθη τότε αυτό το πρόβλημα και αυτό το κείμενο μπορεί να το αναζητήσει κανείς ως υπόδειγμα. Θέματα αυτονομία προπολογισμού. Είναι σύνηθε στα διεθνή δικαστήρια να Καταρτίσουν μόνα τους τον προϋπολογισμό τους και αυτός ο προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει προσφυγή σε άλλες διοικήσεις, σε άλλα διοικητικά όργανα, σε άλλους φορείς όπως η Υπουργική Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και επομένως κανένας τρίτος, όπως παραγματικά ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει σε ουσιαστικό επίπεδο τον προϋπολογισμό μέχρι ότου το τελικό όργανο απόφασης, η Επιτροπή Υπουργών παίρνει μια απόφαση. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να παίρνει το ΕΔΑΔ όλα αυτά τα οποία ζητάει σε επίπεδο προϋπολογισμού. Απλώς λέω ότι το Ευρωπαϊκό το Δικαστήριο, το ΕΔΑΔ και η Επιτροπή των Υπουργών θα πρέπει να βρίσκονται σε ίσο επίπεδο και θα μπορούν να διαπραγματεύονται μεταξύ τους χωρίς παρέμβαση τρίτων. Στην περίπτωση αυτή το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να ε, εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο και το έχει κάνει για το αν οι αιτήσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε διερμηνήσει μεταφραστέ, παραδείγματο χάρη, ήταν πράγματι τεκμηριωμένε ή όχι. Και ζήτησε έγγραφα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί χρειαζόταν αυτοί οι πρόσθετοι μεταφραστέ και διερμηνεί. Και μόνο σε αυτή την περίπτωση επίστη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν υπήρχαν τα τεκμηριωμένα αυτά επιχειρήματα ότι χρειαζόταν πράγματι να θεσπιστούν πρόσθετες θέσεις γλωσσομαθών και νομομαθών. Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι για το καθεστώς των δικαστών στο ΕΔΑΔ. Είναι ουσιαστικά απίστευτο αυτό το οποίο επέβαλε στους δικαστές το Συμβούλιο της Ευρώπης το 89. Υπήρχε μία θητεία η οποία, ε, μάλλον υπήρχε μια θητεία η οποια συνοδευόταν από μια αποζημίωση η οποία μειωνόταν κατά 10% αν ήταν τρεις μέρες άρρωστος ο δικαστής και πολύ περισσότερο στα 50% αν η ασθένειά του περνούσε ένα χρονικό διάστημα. Αυτό για τους αρχικούς δικαστές. Για τους νέους δικαστές τώρα υπάρχει μια ρύθμιση η οποία τους επιτρέπει να υπάρχει μια σύνταξη επί τη βάση των αποδοχών τους. Όλα αυτά δημιουργούν μια κάποια δυναμική, δηλαδή βελτιώνουν το καθεστώς των δικαστών, το καθεστώς του δικαστηρίου και στη δήλωση του Interlagen υπάρχει μια πρόσθετη παράγραφος η οποία έχει προσαρτηθεί, η οποία αποδίδει και μια συγκεκριμένη ανεξαρτησία στο δικαστήριο από την άποψη αυτή εγώ νομίζω ότι έχει ανοίξει μια χαραμάδα, λιγάκι έχει ανοίξει η πόρτα για την καλύτερη αυτή βελτίωση του καθεστώ των βουλευτών, των ε, δικαστών, συγγνώμη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη μικρή χαραμάδα για να εξασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία των δικαστών, διότι μόνο σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει μια απόλυτη ανεξαρτησία των δικαστών. Μόνο οι δικαστέ οι οποίοι δεν έχουν δει διοικητικά εμπόδια και δυσκολίες μπορούν να εκπληρώνουν το λειτουργήμά τους με πλήρη ανεξαρτησία και αυτό είναι απαραίτητο να το εξασφαλίσουμε. Ευχαριστώ. E σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρίβεια των ε, λεκθέντων σας. Και τώρα παρακαλώ να μας μιλήσει ο καθηγητής Ζαν Πολ Ζακέ καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στασβουργού και επίτιμος Γενικός Διευθυντής ε, του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να απαντήσω σε ένα ερώτημα που θέσατε. Γιατί η προσχώρηση δεν αλλάζει τι αρμοδιότητε τη Ένωση και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει απλά, παίρνω παράδειγμα, ότι τότε η Ένωση οφείλει να τηρεί τη θρησκευτική ελευθερία αυτό δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να ψηφίσει κανονισμό ή οδηγία για την ελευθερία του θρησκεύματος. Το γεγονός ότι σέβεται αυτό το δικαίωμα δεν της δίνει το δικαίωμα να νομοθετεί σε όλα τα θέματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει προσχώρηση στην σύμβαση. Σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Βετρανός συνάδελφο έθεσε ένα ερώτημα. Τα εθνικά κοινοβούλια φροντίζουν να υπάρχει σεβασμός των ε, δικαιωμάτων της σύμβασης. Γιατί να, Γιατί γίνει προσχώρηση. Διότι, πρώτον, υπάρχουν πράξεις που προέρχονται από την Ένωση χωρίς εθνική παρέμβαση, όπως οι κανονισμοί, κοινωτικοί κανονισμοί εννοώ. Εκεί σε αυτά κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεύτερον, για οτιδήποτε θέμα που αφορά το κοινοτικό δίκαιο, την τελική απόφαση την έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όχι τα εθνικά δικαστήρια. Συνεπώ έχουμε πράξεις της Ένωσης για τις οποίες μπορεί να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο κλπ. Τώρα έρχομαι επί τη ουσία σύντομα. Άλλοι ομιλητέ ήδη το είπανε. Η Ένωση ήδη εφαρμόζεται τη σύμβαση. Τι νόημα έχει η προσχώρηση. Γενικέ αρχέ με βάση το άρθρο 6, ελάχιστε προδιαγραφέ με βάση τη χάρτα. Αυτό που προσθέτει η προσχώρηση είναι. Το δικαίωμα προσφυγής των ατόμων. Οι πολίτες μπορούν να κάνουν προσφυγή κατά μια πράξη Ένωση που να ελέγχεται από ένα εξωτερικό όργανο τη Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ένωση υπόκειται στο ίδιο καθεστώ με τα κράτη-μέλη, υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο. Αυτό θα είναι το νέο στοιχείο του συστήματο. Για να απαντήσω στο ερώτημα του εισηγητή. Διαπραγματεύσει. Φυσικά τι κάνει η Κομισιόν. Η συνθήκη δίνει στην Κομισιόν το μονοπόλιο τη εξωτερική εκπροσώπηση. Αν υπάρχει εντολή που τη δέχονται τα κράτη-μέλη στις διαπραγματεύσεις, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από την εντολή αυτή. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης, συνεπώς, δεν μπορούν να έχουν λέγην εξ ονόματός τους. Αυτά όσον αφορά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Μία συμβολή. Κατά τη γνώμη μου, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να μείνουν μόνο στα πλαίσια του του αναγκαία, γιατί το να αλλάζουμε την ε, σύμβαση με διάφορες επιπλέον φανταστικές, θα έλεγα, φανταστικού χαρακτήρα δηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σπατάλι χρόνο. Όλες οι άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης θα πρέπει να τις πιστούν. Αν θέλουμε οι διαπραγματεύσεις να κρατήσουν αιώνε, μπορούμε να το κάνουμε. Αν όχι, εγώ θα έλεγα να μείνουμε στα άμεσα και να μην αλλάζουμε τη σύμβαση παρά μόνο στο ότι χρειάζεται για την προσχώρηση. Διαφορετικά θα βασιλεύσει η αδιαφορία. Δεύτερον, ποιο πεδίο πρέπει να καλύπτει η σύμβαση. Σε τι ισχύει η σύμβαση. Η προσχώρηση συγκεκριμένα της σύμβασης. Προσχώρηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτό καινούριο. Σε ποιο πρωτόκολλο πρέπει να γίνει προσχώρηση. Εγώ δεν λέω όχι προσχώρηση, δεν λέω προσχώρηση σε αυτά που θα πρέπει, τα πρωτόκολλα πρέπει να δεκτούν τα κράτη-μέλη και μένουν. Διότι η Ένωση έχει διαφορετική νομική προσωπικότητα από τα κράτη-μέλη. Διότι αν η Ένωση επικυρώσει ένα πρωτόκολλο, αυτό το πρωτόκολλο ισχύει για την Ένωση και δεν ισχύει για τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις εθνικές τους αρμοδιότητες, αυστηρά εθνικές. Το γεγονός ότι το ΕΒ δεν επικύρωσε ένα πρωτόκολλο θα παραμείνει μη επικύρωση, ως μη επικύρωση του πρωτοκόλλου. Δεν θα ισχύει αυτό για τα καθαρά εσωτερικά βρετανικά θέματα. Έπειτα, το κριτήριο μου δεν είναι οι αρμοδιότητες της Ένωσης. Θα ήταν λάθος αυτό. Όχι επειδή δεν υπάρχουν αρμοδιότητες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα τομέα. Παίρνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τη δουλειά του εισηγητή. Το πρωτόκολλο για τη θυματική ποινή που αποκλείεται. Αυτό δεν γίνεται επειδή η Ένωση δεν θα επιβάλλει τη θανατική ποινή και γι' αυτό δεν πρέπει να επικυρώσει το πρωτόκολλο. Δέτε τη συμφωνία έκδοση μεταξύ Ένωση και ΗΠΑ. Τι λέει αυτή η συμφωνία. Έχει μια ρήτρα με βάση την οποία δεν γίνεται Έκδοση όταν κάποιο διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί τη θανατική ποινή στι ΗΠΑ. Άρα υπάρχει σεβασμό τη απαγόρευση τη θανατική ποινή. Ο φίλο ε, Μεντεστεβίγκου το θυμάται. Υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μια αρμοδιότητα να κάνει κανεί κάτι και την υποχρέωση να σεβαστεί ένα δικαίωμα. Άλλο παράδειγμα. Όταν εγκρίθηκε ένας γεωργικός κανονισμός για τη μέθοδο σφαγής των ζώων στα σφαγεία δεν υπήρχαν αρμοδιότητα για την ελευθερία του θρησκεύματος, αλλά διαπιστώθηκε ότι αν δεν προβλεπότερα μια εξαίρεση για τον τελειτουργικό τρόπο σφαγής, θα είχαμε παραβίαση της ελευθερίας του θρησκεύματος. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει προσχώρηση σε όλα τα πρωτόκολλα, όπως είπε ο φίλος Αντώνιο, τα οποία αναφέρονται σε ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία υπάρχει εγγύηση από, το, από τη χάρτα. επειδή η προσχώρηση φέρνει στο φως αρνητικές τάσεις και ας θυμηθούμε τι έγινε με την συνθήκη ξύ, τεχνικά ξαναξυπνάνε ορισμένα επιχειρήματα που ήταν εχθρικά παλιότερα στην προσχώρηση λένε επιχειρήμα που λένε να αποκλειστούν τα πρωτογενή δικαιώματα δηλαδή το δικηστήριο του Στρασβούργου δεν πρέπει να ελέγχει τις συνθήκες είναι διασκεδαστικό αυτό θα μπορούσε και η Γερμανία να αποκλείσει το θεμελιώδες δίκαιο της χώρας. Μα κάθε χώρα υπόκειται στον έλεγχο του συντάγματος. Γιατί να το αποφύγει αυτό η Ένωση, να θέλει να το αποφύγει. Έπειτα, εν πάση περιπτώσει, οι συνθήκες δεν είναι πράξεις της Ένωσης, είναι πράξεις των κρατών μελών και μπορεί να γίνει προσφυγή κατά του κάθε κράτους μέλους ατομικά ή συλλογικά για παραβίαση. Άλλο επιχείρημα. Στην ε, καταμερισμό αρμοδιοτήτων εσωτερικών της Ένωσης. Αυτό είναι καθαρά εσωτερικό εθνικό θέμα. Το Στρασβούργο δεν θα πρέπει να αποφασίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των Βρυξελών. Ο βασικός κανόνας είναι να επιτρέψουμε τους πολίτες, τα άτομα, να κάνουν προσφυγή κατά κράτους μέλους ή κατά της Ένωσης και η Ένωση αν κρίνει ότι υπάρχει θέμα αρμοδιότητας με δική της πρωτοβουλία να περάσει στη θέση της υπεράσπισης. Δηλαδή αν ε, θεωρήσει ότι υπάρχει πρόβλημα κοινωτικού δικαίου να προσφύγει στο δικαστήριο η Ένωση. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, υπάρχουν πολλά αισθήματα, ο Λιβιέτα ανάφερε αλλά όχι το σύστημα Βόσφορος, όπου η Ιρλανδία υπέστη προσφυγή για μια πράξη της Ένωσης και η Ιρλανδία υπεράσπιζε την Ένωση. Πού είναι η δικαιοσύνη εδώ, πού είναι τα δικαιοσύνη. Όταν ε, ε, γίνεται προσφυγή κατά της Ένωσης, δεν θα πρέπει η Ένωση να περιμένει να την υποστηρίξει η Μάλτα ή ένα άλλο κράτος μέλος η καταδίκη είναι αλληλέγγυη. Κατά κάποιο τρόπο καταδικάζεται και το κράτο μέλο και η Ένωση και μετά στα μεταξύ του. Και αν δεν είναι ικανοποιημένοι, α πάνε στο Λουξεμβούργο να λυθεί το θέμα των αρμοδιοτήτων. Άλλο θέμα, πολύ σοβαρό, είναι το θέμα του μονοπωλίου της ερμηνείας του δικαστηρίου. Το δικό μας δικαστήριο που έχει το μονοπόλιο ερμηνείας του δικαίου της Ένωσης και μας λένε ότι το Στρασβούργο θα ερμηνεύσει το δίκαιο της Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε την εξή αρχή. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είπε ότι δεν ερμηνεύει το εθνικό δίκαιο. Έτσι λοιπόν δεν ερμηνεύει το δίκαιο της Ένωσης. Αυτό είναι γεγονός για το δικαστήριο το βλέπει ως έχει το δίκαιο. Αν το έκανε και αν το έκανε με κακό τρόπο, αν έκανε λάθος, ε, θυμηθείτε ότι στη συνέχεια οι αρχές της Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να πούνε ερμηνεύσαμε λανθασμένα το δικαιό μας, ε, κάναμε λάθος, ε, γιατί εμείς είπαμε ότι το δικαιό μας θέλει να πει αυτό το οποίο συνάδει με τη σύμβαση. Και έτσι λοιπόν θα υπάρξει διόρθωση. Όμως αυτό θα γίνει αφού έχουν εξαντληθεί τα, εθνικά ένδικα μέσα. Αν ε, υπάρχει άμεση προσφυγή ενός ε, πολίτη στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, πρέπει πρώτα να πάει να προσφύγει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου και κατόπιν στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Αν ε, εμφανιστεί ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου, Νομίζω ότι είναι απλό το σύστημα, έχει την υποχρέωση ε, σύμφωνα με την ΕΣΔΑ να ζητήσει προδικαστική παραπομπή στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Γι' αυτό είναι θέμα δικαίου της Ένωσης. Αν δεν το έχει κάνει, δεν έχει εξαντλήσει τα ε, εσωτερικά ενδικά μέσα και αν το κάνει και το Εθνικό Δικαστήριο πει όχι. Αν ε, είναι θέμα εγκυρότητας καταρχήν παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης η ε, νομολογία υποχρεώνει ε, να, να εξεταστεί το θέμα της εγκυρότητας και δεν υποχρεώνει την υποχρεωτική προσφυγή στο Λουξεμβούργο. Όμω αυτό δεν ισχύει σε όλε τι περιπτώσει. Αν ο δικαστή δεν δώσει συνέχεια στην προσφυγή, δεν ε, έχει παραβιάσει στο δικαίωμα της ισότιμης δίκης. Και αν πάμε στο Στρασβούργο και ε, πείτε Στρασβούργο δεν θέλω να εξετάσω την υπόθεση επί αλλά διαπιστώνω ότι δεν ε, χρησιμοποιήσετε την προδικαστική ε, παραπομπή, έτσι λοιπόν παραβιάστε την διαδικασία. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πολλά στοιχεία της νομολογίας ε, του Δικαστηρίου του Στρασβούργου που πρέπει να δούμε. Έτσι λοιπόν ίσως θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε ποια είναι τα εσωτερικά ενδικά μέσα. Τώρα για την προσφυγή. Είναι προφανέ ότι αποκλείεται η προσφυγή μεταξύ κρατών μελών. Ε, ναι, για την προσφυγή τρίτων κρατών. Να πω ότι η Ρωσία έχει επικυρώσει το πρωτόκολλο 14. Έτσι λοιπόν ε, επιτρέπεται η προσχώρηση της ε, Ένωσης. Ε, έτσι νομίζω τώρα ότι πρέπει να απλοποιούμε τα πράγματα, να μην αφευρίσκουμε συστήματα όπου ο πολίτης θα πρέπει να κάνει μια προσφυγή στο Λουξεμβούργο που θέτει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Στρασβούργο κτλ. Αν θέλετε μια δίκη που θα κοστίσει ακριβά και θα κοστίσει και 20 χρόνια, μάλλον αυτή είναι η καλύτερη οδός. Ο πολίτης θα πρέπει να κρίνει ποιο είναι το συμφέρον του αν κρίνει ότι δεν αξίζει τον κόπο και θα κοστίσει ακριβά, δεν θα πάει στο Στρασβούργο. Ο πολίτης πρέπει να είναι ελεύθερος για την επιλογή του, για να επιτελέσει την επιλογή του. Τώρα για το θέμα της συμμετοχής. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρώτο θέμα διαπραγμάτευσης. Ε, ε, πηγαίνουμε, λέμε ότι θέλουμε πλήρη συμμετοχή. Θα έχουμε και το δικαστή και την Επιτροπή που θα ψηφίζει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Δικαιωμάτων. Ε, διαφορετικά μπορούμε να πούμε όχι δεν θέλουμε τα πάντα. Και λέω στο εγγραφό μου ότι υπάρχουν και θέσεις αναδίπλωσης και θα κλείσω, Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Η προσχώρηση δίνει στον ιδιώτη, αποκαθιστά στον ιδιώτη, είναι δικαίωμα που το είχε κλαπεί. Πριν ε, να μεταφερθεί η αρμοδιότητα από τα κράτη-μέλη στην Ένωση, όταν τα κράτη-μέλη είχαν αρμοδιότητα στα γεωργικά θέματα, μπορούσε ο ιδιώτης να προσφύγει στο Στρασβούργο για να παραπονεθεί για μία νομοθεσία για τον τομέα της γεωργίας. Ενώ σήμερα δεν μπορεί να το κάνει γιατί την αρμοδιότητα για τα γεωργικά την έχει Ένωση και δεν ε, έχει προσχωρήσει. Έτσι λοιπόν, ε, τελικά τι λέει εδώ ο πολίτης, επιστρέψτε μου το δικαίωμα που μου έχει κλέψει η Ένωση. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Και τώρα θα έχουμε την ε, τρίτη παρέμβαση του καθηγητή Ολιβιέντε Σούτερ, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν Λανέβ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια μεγάλη ε, ευχαρίστηση και μια πρόκληση να λαμβάνω το λόγο μετά από τον Ζω Πολ Ζακέ. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα από τα σημεία που παρουσιάστηκαν στη συζήτηση χωρίς να επαναλάβω, ελπίζω, αυτά που ελέγχθηκαν. Θα σταθώ σε τέσσερα σημεία, τα οποία είναι σημεία τα οποία έχω αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό, σε ένα υπόμνημα, το οποίο σας έδωσαν, ελπίζω, χθε οι υπηρεσίες της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα, η περίφημη αυτή αρχή της αυτονομίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που βρίσκεται στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αναφέρεται στα άρθρα 19 παράγραφος 1 και 344 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή σημαίνει κάτι το πολύ απλό, ότι τα θέματα ερμηνείας και εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να υπόκεινται στον τελικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έχει το μονοπόλιο ερμηνείας νομικής του κοινοτικού δικαίου. Από την αρχή αυτή απορρέουν δύο συνέπειες. Πρώτα απ' όλα, δεν εναπόκειται στο ΕΔΑΔ να αποφασίσει ποιες είναι οι αρμοδιότητες, οι αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, Αντίθετα, να στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη να καθορίσουν αυτή την κατανομή αρμοδιοτήτων μόνοι τους υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι θεμητή αυτή η ανησυχία η οποία εκφράζεται πολλές φορές και η οποία λέει ότι το να υποκείμεθα στον έλεγχο του ΕΔΑΔ, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ανατραπεί και η ισορροπία των αρμοδιοτήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι η καλύτερη πρόσφορη λύση θα είναι να δώσουμε σε οποιοδήποτε κράτο μέλος, το οποίο είναι υπόλογο για οποιοδήποτε μέτρο το οποίο έχει λάβει, να είναι υπόλογο και ενώπιον του ΕΔΑΔ και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα να εγκαλείται ένα κράτος μέλος όπως γίνεται στις αστικές δίκες μέσω της ε, επιτακτικής παρέμβασης, της αναγκαστικής παρέμβασης. Αυτό σημαίνει ότι δίδεται η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολιτέ και στα κράτη-μέλη όταν παρουσιάζεται μία υπόθεση στο ΕΔΑΔ που αφορά ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα κράτος μέλος που εμπλέκει την δική της αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ένας μηχανισμός αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το σχέδιο ψηφίσματο νομίζω ότι αναφέρει εδώ σε αυτήν την περίπτωση που λέει ότι εναπόκειται στο ΕΔΑΔ ή στην Προεδρία του ΕΔΑΔ να δώσει την έγκρισή του για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι αυτεπάγγελτη αυτή η δυνατότητα παρέμβασης, γιατί μπορούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ΕΔΑΔ θα μπορούσε να έχει κάποια προκατάληψη σε ό,τι αφορά την εσωτερική κατανομή ισορροπίας εξουσιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Η παρέμβαση αυτή δεν θα γίνεται από θεσμικούς φίλους μέσα σε εισαγωγικά όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να παρέμβει, αλλά από αυτούς οι οποίοι έχουν ένδικο συμφέρον και θα έχει εκτελεστό χαρακτήρα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό υλοποιεί επομένως την ιδέα της αλληλέγγυας και κοινή ευθύνη. Οι μηχανισμοί τώρα αυτοί θα έχουν σαν αποτέλεσμα πρώτον ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε μια συμφωνία για ένα κατάλογο αρμοδιοτήτων, κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο να το κάνουμε με εξαντλητική απαρίθμηση, διότι αυτό οι αρμοδιότητε μεταξύ των μελών και Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσονται συνέχεια σε ό,τι αφορά την ισορροπία του. Δεύτερον, δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να καθορίσουμε τι ευθύνε των μεν και των δε πριν από την απόφαση του ΕΔΑΔ. Τέσσερα-πέντε χρόνια διαρκεί μια διαδικασία στο ΕΔΑΔ, όπω ξέρετε, κατά μέσον όρο. Και αν προσθέσουμε ένα μηχανισμό καθορισμού αρμοδιοτήτων μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πρέπει να γίνει αυτό απριόρι, αυτό θα επιμηκύνει ακόμα με τρόπο παράλογο τη διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑ. Τρίτον, πιστεύω ότι ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μια συμφωνία μεταξύ τους σε σχέση με τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του ΕΔΑΤ, βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να πριτανεύει όπως λέει και το άρθρο 4 παραγωγός 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δεύτερη απόρρια της αρχής της αυτονομίας είναι ότι αποκλείονται οι οριζόντιοι μηχανισμού ελέγχου μέσα στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή οι διακρατικές προσφυγέ όπω αναφέρεται στο άρθρο 33 τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν προσφυγέ έναντι αλλήλων όταν πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ίσως ρευστό και δύσκολο το σύνορο μεταξύ των δύο για να το καθορίσουμε, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε απόλυτα βάσει του άρθρου 33 τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τι προσφυγέ μεταξύ κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν να κάνουν το κοινοτικό δίκαιο. Δεν είναι μια αποσύνδεση κατά κάποιο τρόπο από το δικαστή των κρατών μελών που τα απαλλάσσει από τον έλεγχο τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά θα είναι μια τέτοια ειδική ρύθμιση που αναφέρεται ήδη στο άρθρο 55 της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που λέει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν μεταξύ τους να προβούν σε συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ των οποίων αποφασίζουν να μην προσφεύγουν εναντίον αλλήλων ή να μην ε, υποβάλλουν στο ΕΔΑΔ ε, υποθέσεις οι οποίες έχουν αποφασίσει να τις επιλύουν με άλλο τρόπο. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να τονίσω είναι οι δύσκολες αυτές καταστάσεις όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου δεν είναι σε θέση να αποφανθεί για ένα θέμα που έχει να κάνει με συμβατότητα με την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προτού αυτό εξεταστεί από το ΕΔΑΤ. Αυτό είναι μια πραγματική δυσκολία. Δεν είναι μονάχα στι Βρυξέλλε αλλά και στο Λουξεμβούργο, που πολλέ φορέ υπάρχουν ερωτήματα τα οποία οδηγούν σε νευρικότητα και δυσκολίε. Υπάρχουν καταρχήν καταστάσεις, οποίες αναφέρει και ο Ζωάν Πολ Ζακέ, όπου η τωρινή συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζει την αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του απαγορεύει να εκφέρει απόψη και να αποφασίσει για ορισμένα θέματα, τα οποία παρόλα αυτά προκύπτουν από μέτρα που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι η περίπτωση της ΚΕΠΑ, το άρθρο 215 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει σε οριακέ περιπτώσει μια αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά όχι σε όλε τι περιπτώσει. Ή αν δούμε το άρθρο 276 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο σε σχέση με το χώρο δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, λέει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα για να ελέγξει την εγκυρότητα και την αναλογικότητα ενεργειών που έχουν να κάνουν με θέματα αστυνομικά, ασφάλεια και δεν πρόκειται να παριθμίσει όλε τι πτυχέ αυτού του άρθρου. Σε τέτοιου είδου περιπτώσει είναι τροτό το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τροτό διότι αυτό οφείλεται στη θέληση των συντακτών των συνθηκών που είναι τα κράτη-μέλη, που θέλησαν καταρχήν εν μέρη να απαλλάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ε, έλεγχο του δικαίου, αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε αν είναι πράγματι συμβατό με το άρθρο 13 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που δεν προβλέπει καμία εξαίρεση από αυτό τον έλεγχο το δικαστικό. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι υπάρχει μια συμπληρωματικότητα η οποία πρέπει να υπάρχει μεταξύ των εθνικών ειδικών μέσων που οργανώνονται από τα κράτη-μέλη και της πρόσβασης στο ΕΔΑΔ, μάλλον της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί αναφέρει συνθήκη στο άρθρο 19 ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρξει αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος στον τομέα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι έλκεται και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τα κράτη-μέλη θα πρέπει με την οργάνωση εθνικών ενδίκων μέτρων να καλύψουν και να συμπληρώσουν την πολλές φορές ανεπαρκή προστασία που δίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω των ορίων που υπάρχουν για την αρμοδιότητα αυτού του δικαστηρίου. Μια άλλη κατάσταση είναι αυτή στην οποία αναφέρθηκε και πάλι ο κύριος Ζακέ, έχει να κάνει με το ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν σέβονται τις υποχρεώσεις τους, δεν κάνουν τη δουλειά τους, να θέσουν προδικαστικό ερώτημα για την ε, ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο 10 κατά παραβίαση του άρθρου 276 της συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει από τις αρχές μια υποχρέωση. Θεωρώ ότι ακόμα και αν το ε, ΕΔΑ δεν το έχει πει ρητός ότι ο εναγων, ενώπιον, μίας, ενώπιον ενός δικαστή ε, στο ΔΕΚ δεν έχει εξαντλήσει όλα τα εθνικά ένδικα μέσα όπως θα έπρεπε να κάνει, ε, τότε αν προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου η αγωγή του θα ε, κηρυχθεί απαράδεκτη. Η προσφυγή του θα κηρυχθεί απαράδεκτη. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε αυτή τη βεβαιότητα ότι ε, θα υπάρχει προσφυγή στο δικαστήριο του Στρασβούργου πάντοτε αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα εθνικά ένδικα μέσα. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτό θα πρέπει να το καθορίσει το δικαστήριο του Στρασβούργου δυνάμει του άρθρου 13 της ε, σύμβασης της ΕΣΔΑ. Λοιπόν, για να μείνω και στα πλαίσια του χρόνου, δικαίωμα ψηφοφορία, δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή των Υπουργών θα τεθεί το ερώτημα αν θα πρέπει γι' αυτό να τροποποιηθεί το καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, το σχετικό άρθρο που προβλέπει, τον τρόπο ψηφοφορία στην Επιτροπή των Υπουργών. να είναι η απάντηση είναι θετική, τότε το εμπόδιο δεν θα είναι οπότε όπως και να έχει πράξη προσχώρησης, ε, θα κυρωθεί από τα 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να γίνει μια τροποποίηση στο καταστατικό επί αυτού του συγκεκριμένου σημείου. Εγώ νομίζω όμως ότι ότι ένα ψήφισμα τη Επιτροπή των Υπουργών θα μπορούσε να αρκέσει. όμω το σχέδιο έκθεση που μα υποβάλλεται υπάρχει ένα τεκμήριο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια πρόσθετη ψήφο που θα προσθεθεί κατά κάποιο τρόπο στις 27 ψήφους των κρατών μελών. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε κακόπιστοι, κάθε κράτος μέλος τη Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχε 1,37 ψήφους στην Επιτροπή των Υπουργών, γιατί τελικά εκπροσωπείται δύο φορές και από τον εαυτό του και μέσω της ε, ψήφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι η προσθήκη μιας προσθέτης ψήφου θα σύναδε με την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος, αλλά αυτό μπορεί μπορεί να προκαλέσει κάποιο εκνευρισμό και ούτω ή άλλω μπορεί να θεωρηθεί κάτι συμβολικό. Μία εναλλακτική είναι η αλλω μπορει να θεωρηθει κατι συμβολικο Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη από κοινού να διαθέτουν 27 ψήφου στην Επιτροπή των Υπουργών και από κοινού αν ε, θεωρούν ε, ότι το θέμα ε, χρήζει ανάληψη κοινωτικής πρωτοβουλία, θα μπορούν να ασκήσουν αυτή την ψήφο από κοινού. Αυτή τη η λύση έχει επιλεχθεί στο άρθρο 44 των ΗΠΑ για τα άτομα με ανεπηρία. Εκεί προβλέπεται ο τρόπος αυτός άσκησης του δικαιώματος ψήφου. Και θα κλείσω συγχαίροντας τον συγητή για την παράγραφο που αφιέρωσε στο τέλος του σχεδίου ψηφίσματος σε ένα θέμα που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του 1996, τον θεωρημένο χάρτη τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αδιέρετα και πάρα πολύ σημαντικά τα οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά δικαιώματα πρέπει να θεωρούνται τόσο σημαντικά όσο και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο ίδιο η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων το δηλώνει αυτό το θέμα και μέσω μία δομής που ήθελε ουσιαστικά να μην ακολουθήσει την παραδοσιακή οδό και διαπιστώνω ότι όταν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζονται ενώπιον ε, της Επιτροπής των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αυτού τον εξάρτητου φορέα που εποπτεύει επί του σεβασμού των δικαιωμάτων, πολύ συχνά ε, έρχεται να υπερασπιστεί το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της εισαγωγής διακρίσεων, για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την ασφάλεια στην εργασία και θεωρώ ότι είναι φυσικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, χωρίς να υπάρχει υπερβολική καθυστέρηση να δώσει ένα μήνυμα ότι αμελητή ξεκινούμε ένα προβληματισμό για το ο κοινωνικό χάρτη. Αυτό προβλεπόταν και στην συνθήκη Σπινελή που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη έχουμε χάσει 30 χρόνια. Ας μην χάσουμε επιπρόσθετο το χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πράγματι, πάρα πολύ καλά τα πάμε με το χρόνο. Έχουμε σεβαστεί τις προθεσμίες. Θα, ε, ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Μέσα Συγκλητή να έρθει εδώ να με αντικαταστήσει, γιατί πρέπει να λείψω για πέντε λεπτά. Μπορείτε να έρθετε, να προεδρεύσετε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και αρχίζει η, τώρα η φάση της συζήτησης. Πρώτος, ο συνάδελφος Καορέγκουλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε τις τρεις παρεμβάσεις ε, και εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Ζαν Πολζάκ ε, για την ε, σαφήνεια των επιχειρημάτων του και θα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεσούτερ ιδιαιτέρως. Αναφέρθηκε στην ε, ε, παράγραφο 13 της εκθεσής μου και τον ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλα τα μέλη ε, εδώ αυτού του οίκου θα δεκτούν αυτήν την τόσορτη αναφορά στη Χάρτα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολεμική ε, δυστυχώς ε, στο εσωτερικό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν ε, κάποιοι δισταγμοί σε ορισμένες χώρες για την ενσωμάτωση αυτής της έννοιας των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των κοινωνικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με συγχωρείτε, και Επίσης ε, το να ε, έχει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοινωνικό και εργασιακό τομέα. Ε, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αναφορά που κάνατε στην αναγκαιότητα να σκεφτούμε αυτό το θέμα. Η παράγραφος 13 της έκθεσης, όπως είπατε, στέλνει ένα μήνυμα σε σχέση με την αναγκαιότητα να σκεφτούμε επί της κοινωνικής χάρτας στο πλαίσιο μιας τόσο σημαντικής πολιτικής απόφασης όπως είναι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ΕΣΔΑ. Μια ερώτηση έχω ακόμα να υποβάλω. Εσείς πιστεύετε ότι η αναγκαιότητα να διασφαλίσουμε ε, το ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη θα είναι διάδικη σε όλες τις διαδικασίες, ε, επιζητεί, επιφέρει την μεταρρύθμιση του άρθρου 36 της συνθήκης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση αυτή Ε, θα έχει τις απαραίτητες εγγύσεις για να είναι πάντοτε συνεναγόμενοι. Πέρα από ότι το άρθρο 36 δεν αναφέρει τόσο αυτή τη δυνατότητα, θα έπρεπε να γίνει τροποποίηση αυτού του άρθρου της συνθήκης, της σύμβαση Με συγχωρείτε, αυτή είναι η ερώτησή μου. Äh, Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Ευχαριστώ πολύ. Όταν προσυπογράψουμε την ε, σύμβαση, ξέρουμε ότι αυτή θα γίνει πράγματι ένα ουσιαστικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικαίου, παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο του, της Ευρώπης έχει την ουσιαστική αρμοδιότητα και θα είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει αυτή τη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει τη δικαίωση τη δικαιοδοσία να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει δύο διαφορετικά έγγραφα. Την δική του σύμβαση, τη σύμβαση του, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών ρώτησα τον καθηγητή Ζακέ τι θα γινόταν σε επίπεδο ιεράρχηση των δύο εγγράφων. Αν υπήρχε μία σύγκρουση μεταξύ των δύο εγγράφων, ποιο υπερέχει σε νομικό επίπεδο και ελπίζω ότι δεν έχω κάνει λάθο σε αυτό το οποίο μεταφέρω. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι το έγγραφο το οποίο δίνει την ευρύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να έχει υπεροχή ενώ αυτού που δίνει τη μικρότερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά κάθισα και σκέφτηκα και είπα, α υποθέσουμε ότι έχουμε μια περίπτωση δύο διαδίκων που ο καθένα ε, διεκδικεί δικαιώματα τα οποία είναι ασύμβατα μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι κάτι απόλυτα θεωρητικό. Αν πάρουμε την περίπτωση των γελιογραφιών του προφήτη στη Δανία, αυτό είναι μια περίπτωση η οποία θα μπορούσε να προκύψει και στην πράξη. Σε ποιο σημείο το κάθε δικαίωμα, σε κάθε ένα από τα έγγραφα, υπέρεχει του, των αντιστοίχων δικαιωμάτων στο άλλο έγγραφο. Επίσης, τον καθηγητή κ. Σλούτερ, ελπίζω ότι κατάλαβα καλά, γιατί είπατε σε κάποιο σημείο είπατε σε κάποια περίπτωση ότι θα πρέπει να αποκλειστεί η περίπτωση στα κράτη-μέλη να ενάγουν τα μεν τα δε. Δεν ξέρω αν εννοούσατε αν θα πρέπει να αποκλείονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή μόνο από το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Αν γινόταν κάτι τέτοιο, τότε τα κράτη-μέλη θα παρακάμπτανε το Λουξεμβούργο και θα πηγαίνανε μονάχα στο Στρασβούργο. Αν αυτό που είπατε είναι ότι πρέπει να αποκλείονται από προσφυγή στο Στρασβούργο, αυτό όμως θα έπρεπε να αποφασιστεί από το Δικαστήριο από τα κράτη-μέλη να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως όπως η προσφυγή της Ιρλανδίας εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου για τα δικαιώματα των υπόπτων του Ήρα το 1972 αν θυμάμαι καλά. Allora, alla parola... Ο Σεβερίν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, κύριε καθηγητέ για τις παρατηρήσεις σας. Είναι σαφές ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ένωση έχει νομική προσωπικότητα, συνεπώς έχει τη δυνατότητα να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑΡ. Και δεύτερον, υπάρχει απόφαση στη συνθήκη της Λισαβόνας ότι η Ένωση θα το κάνει. Ξεκινώντας από αυτό, θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο και των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Απλώς εκρίθη σκόπιμο να επεκταθεί ο έλεγχος αποφάσεων της Ένωσης όχι μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου αλλά μέσω του Ευρωπαϊκού Συγκρατήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Έτσι, έχουμε εμβάθυνση στην ευρωπαϊκή ενοποίηση για να χρησιμοποιήσουμε μια ορολογία που σε μερικού δεν είναι πολύ δημοφιλής να αυξηθεί ο ομοσπονδιακός χαρακτήρας της Ένωσης. Από αυτή τη σκοπιά, αν δούμε τα πράγματα, δεν θα πρέπει να λυπόμαστε για το ότι το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει ορισμένε περιπτώσει, αλλά να πούμε όχι, αυτό θέλαμε. Θέλαμε και ένα άλλο δικαστήριο, το δικαστήριο του Στρασβούργου, τώρα να μπορεί να ερευνήσει θέματα που, είναι πέραν, που ήταν πέραν δικαστηριακού ελέγχου στο παρελθόν. Δεύτερο, προσχωρώντας ε, στην ε, σύμβαση, κατά κάποιο τρόπο διευρύνουμε το κοινό χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Αυτό είναι ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Κατά κάποιο τρόπο ευρεώνουμε τον δικαστηριακό έλεγχο των αποφάσεων της Ένωσης και δίνουμε πρόσβαση σε αυτού του είδους τον έλεγχο σε αυτούς που δεν ανήκουν σε μέλη της Ένωσης. Και όπως υπόθηκε και συμφωνώ, δίνουν καλύτερη προστασία στους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τα δικαιώματά τους, διότι όσοι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούσαν να προσπίσουν όλα αυτά τα δικαιώματά τους πριν, πριν η Ένωση υπογράψει την σύμβαση. Ένα άλλο σημείο που το θέτω ως ερώτηση οι πολίτες της Ένωσης κρατών που δεν είναι μέλη έχουν δικαίωμα ανεξάρτητης πρόσβασης στο δικαστήριο σε σχέση με αποφάσεις της Ένωσης. Στο ερώτημα αυτό εγώ απαντάω ναι. Άρα δεν είναι ερώτηση, είναι περισσότερο ένα είδος ε, σχόλιο που κάνω για να το αντισχολιάσετε από τη μεριά σας. συμφωνώ με τη γνώμη του καθηγητή Ζακ ότι με τα επιπλέον πρωτόκολλα ουσιαστικά δεν έχουμε προβλήματα. Είναι ένα κακό στερούμενο επίδικο θέμα. Μερικές χώρες μέλη υπέγραψαν μερικά, ή όλα, αλλά όλοι, όλοι είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και με αυτή τους την ιδιότητα όλα τα κράτη-μέλη έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Συν Ενδεχομένω ορισμένα ή όλα από τα πρωτόκολλα. Αυτό σημαίνει όταν τα συγκεκριμένα αυτά κράτη όταν τους ζητηθεί να έρθουν στο δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα κριθούν με βάση τα πρωτόκολλα που έχουν αναγνωρίσει σε εθνική βάση. Αλλά όταν θα έχουμε περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται ως νομική οντότητα για λογαριασμό της κατά κάποιο τρόπο, τότε μπορεί να απαντήσει σε σχέση με όλα τα πρωτόκολλα χωρίς να επηρεάζει τα δικαιώματα των κρατών που δεν έχουν προσυπογράψει όλα τα επιπλέον πρωτόκολλα. Μην μπερδεύουμε αυτά τα δύο θέματα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Γιατί να ανησυχούμε όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Τώρα για το τελευταίο άρθρο του ψηφίσματος, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε αυτό που υπόθηκε, ότι δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναπτύσσεται και υπάρχει ένα συνεκτικό σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν μπορούμε να το κατακαιρματίζουμε. Αντίθετα θα πρέπει να το κρατάμε ενωμένο, ενωποιημένο. Και ακόμα κι αν η συνθήκη της Λισαβόνας ανέλεγε ότι θα πρέπει να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τις άλλες συνθήκες και συμβάσεις στην καθολική έννοια, στην παγκόσμια έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτές θα πρέπει να είναι τμήμα της εντολής μας να συμπεριληφθούν, να προσυπογραφούν κλπ. Αν δούμε τα πράγματα έτσι, μπορούμε να βρούμε τη νομική βάση που μας χρειάζεται προκειμένου να προσχωρήσουμε και στις άλλες συμβάσεις που αποτελούν το σύμπαν κατά κάποιο τρόπο του ε, νομικού συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σεβαρίν. Ο κύριος Νταφ ζήτησε το λόγο. Πρόεδρο. Όπως είπαν οι υπονόησαν και οι προελελήσαντες ότι θα πρέπει τα πρόσθετα πρωτόκολλα, η σχετική προσχώρηση στα πρόσθετα πρωτόκολλα, θα πρέπει να εξεταστεί ένα περίπτωση. Δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία όπως θα μπορούσε να φανεί εκ πρώτης όψεως. Αλλά θα πρέπει να ελέγξουμε αν συναντούν τα πρωτόκολλα με τη χάρτα και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι ένα εγχείρημα που θα πρέπει να υλοποιήσουμε πριν την υλοποίηση της προσχώρησης. Να ρωτήσω, αυτό το εγχείρημα της προσχώρησης τα πρόσθετα πρωτόκολλα θα πρέπει να γίνει ως τμήμα των διαπραγματεύσεων της προσχώρησης ή μπορεί να αναβληθεί. για το μέλλον. Δεύτερη ερώτηση. Κύριο Σάγγελ, μας ε, περιέγραψε κάπως ζωφερό όλο αυτό το γραφειοκρατικό άχθος ε, που αφορά το δικαστήριο και τη λειτουργία του. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρχει ένα κόστος για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ΕΣΔΑ και φυσικά το κόστος πάντα ενδιαφέρει το Κοινοβούλιο. Μήπως θα μπορούσατε να μας αναφέρετε και κάποια νούμερα, πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με το κόστος. Δεν μου απαντήσατε επίσης και στην προηγούμενη ερώτησή μου. για την ε, κατάλληλη εκπροσώπηση στην Επιτροπή των Υπουργών. συμφωνείτε ότι θα έπρεπε να είναι η Επιτροπή η οποία θα προβαίνει σε αυτήν την εκπροσώπηση. Μέντε, δεν Δεβίγου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη χρειάστηκα να βγω λόγω κάποιου αστάθμητου στοιχείου. Μία από τι ερωτήσει τώρα αν έχει ήδη απαντηθεί, σας ζητώ συγγνώμη. Μπορείτε να την αγνοήσετε. Θέλω να θέσω το θέμα των επιφυλάξεων που μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη ή που παρουσιάσανε για τα πρόσθετα πρωτόκολλα τα οποία, τα οποία συνδυάζονται με την ε, ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρουσιάσει επιφυλάξει. Έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση από εσά. Δεύτερον, κύριε Σεβερίν, θέσατε ένα ζήτημα το οποίο περιλαμβάνεται και στο ψήφισμα του κύριου Άουτ. Χαουρεγγί. Το ψήφισμα αναφέρει στην τελευταία παράγραφο για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη των εμπειρογνωμόνων για το ζήτημα αυτό. E ευχαριστώ. Ο κύριος Πουσουτήλ έχει ζητήσει το λόγο. Yes, thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτής τόσο ενδιαφέρουσας ημερίδας. Συζητήσαμε χθες την γνωμοδότηση της κυρίας Κίνγκα Γκάλ στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Ήταν χθε τη μέση έδεξη το θέμα αυτό και εγώ έθιξα κάτι το οποίο θέλω να το αναφέρω και πάλι σήμερα. Και θα ήθελα ίσως να έχω μια απάντηση από τους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς προσκεκλημένους μας. Πρόκειται για την σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του ΕΔΑΔ, που για μένα είναι πραγματικά συναρπαστική αλλά και πολυδέδαλη. Και εδώ καταγράφω ότι για πρώτη φορά θα έχουμε ένα δικαστή που δεν θα προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος ουσιαστικά θα μπορεί να αποφασίσει για στοιχεία αγκυρότητας του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα δικαστήριο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να αντιμετωπίσει την εγκυρότητα του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω αν αυτό οδηγεί σε κάποιες αντιδράσεις από τους εμπειρογνώμονες. Υπάρχουν προβλήματα παραγωγικά και ερωτήματα για το κατά πόσο άτομα τα οποία δεν έχουν εμπειρία στο να αποφασίζουν θέματα σε σχέση με, την, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εμπλέκονται στην λήψη αποφάσεων για την τελική εγκυρότητα, σε τελική ανάλυση εγκυρότητα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τους εμπειρογνώμονες μας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους ε, προσκεκλημένους μας, ε, τους εμπειρογνώμονες, ποιος θα ήθελε να απαντήσει σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν, ε, ακούσατε τις ερωτήσεις από τους συναδέλφους, ποιος από σας θα ήθελε να απαντήσει. Παρακαλώ. Πρόεδρε, Υπάρχουν ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Ακούσαμε τον κύριο Ντεβίγο ε, για το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, όπως είπε και ο κύριος Ντεσούτερ, να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε στη τη χάρτα και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι πριν ε, να έχουμε 40 βαθμούς ε, τη μέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα, γιατί αυτό το κράτος ε, θέτει πολλά προβλήματα. Αλλά είχαμε και κράτη που ήταν εντελώ αντίθετα στην προσχώρηση και τα καταφέραμε τελικά μετά από 30-40 χρόνια. Έτσι τελικά δεν ξεκινήσουμε από κάπου, τελικά πουθενά δεν θα καταλήξουμε, είναι μια αρχή. Τώρα, για το θέμα του εισηγητή, για την ερώτηση του εισηγητή. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι συναγόμενη ένωση και μην αφήνει τα κρατημέλη να διεκπεραιώνουν τα ζητήματα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε κριτήρια, γιατί αν θέσετε κριτήριο, τότε αυτό θα αφορά απλώς το δίκαιο της Ένωσης και τελικά το δικαστήριο του Στρασβούργου θα αποκτήσει αρμοδιότητα επί της αρμοδιότητας ε, για το δίκαιο της Ένωσης. Ε, στον ε, ΠΟΕ, στην ΚΑΤ, τις έχουμε δει αυτές τις δυνατότητες. Για την εκπροσώπηση στην Επιτροπή των Υπουργών. Ναι, φυσικά. Αυτό θα γίνει μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βλέπω ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουμε, να εγκαταλείψουμε εδώ την κλασική λογική των συνθήκων. Τώρα για τη σχέση μεταξύ των συστημάτων. Να επαναλάβω ότι η σύμβαση ήδη ανήκει στο δίκαιο της Ένωσης. Έτσι δηλαδή όποιο θέμα προβλήματος μεταξύ σύμβασης και χάρτας ειδητήθηκε σήμερα. Τη λύση που, η λύση που βρήκαμε είναι η εξή. Να πούμε όπως προβλέπετε στη χάρτα ότι η σύμβαση αποτελεί ένα ελάχιστο πρότυπο, κάτω από το οποίο δεν μπορεί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορεί να πάει πιο μακριά. Τώρα το πρόβλημα με τα σκίτσια, κοιτάξτε, αν είναι πιο ε, αν προσφέρει μεγαλύτερη προστασία η χάρτα, εφαρμόζουμε τη χάρτα, αν προσφέρει μεγαλύτερη προστασία η σύμβαση, χρησιμοποιούμε τη σύμβαση. Τώρα για το θέμα των δύο δικαστηρίων. Εγώ δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ασυνέπεια. Θα ήθελα όμως να πω ότι δεν κάνουν το ίδιο πράγμα τα δύο δικαστήρια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πλήρη αρμοδιότητα για το δίκαιο της Ένωσης, ενώ το δικαστήριο του Στρασβούργου έχει επικουρική δευτερεύουσα αρμοδιότητα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έτσι λοιπόν, τίποτα δεν αφαιρείται από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, υπό την επιφύλαξη βέβαια ε, ότι ε, έχουμε εκεί το μονοπόλιο της ερμηνείας του δικαίου της Ένωσης, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα συνεχίζει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε πάντα. Αυτό που προσθέτουμε είναι ένα επιπρόσθετος έλεγχος για την ερώτηση τώρα που τέθηκε αν ε, μας ενοχλεί ότι θα έχουμε ε, άτομα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποφαίνονται επί του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ενοχλεί τη Γερμανία, ε, ένας δικαστής Τσέχος από το Στρασβούργο να μπορεί να αποφαίνεται επί θεμάτων που αφορούν την Ένωση. Κοιτάξτε, αν θέλουμε ανεξάρτητη κρίση, πρέπει να έχουμε κάποιους τρίτους που θα κρίνουν. Τώρα, για το πρωτόκολλο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη εφαρμόσει ορισμένα πρωτόκολλα. Το πρωτόκολλο υπεριθμών 1, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ήδη εφαρμόζεται. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει αναθεώρηση. Όλα τα δικαιώματα που καλύπτονται από τη χάρτα θα πρέπει καθολικά να προστατεύονται και από την Ένωση. Ευχαριστώ. να δώσουμε το λόγο και στους ε, άλλους εμπειρογνώμενους, κύριο ε. Θέλετε κάτι να πείτε. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε, λέει ο Τέσσερα σημεία είναι αυτά τα οποία με οδηγούν στο να παρέμβω μεταξύ αυτών που αναφέρθηκαν και νομίζω ότι μπορώ να ακολουθήσω τη σειρά με την οποία αναφέρθηκαν τα θέματα αυτά. Το ερώτημα του κυρίου Χαουρεγή καταρχήν για την θέση του συναγω... συνεναγωμένου που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχει μια προσφυγή εναντίον τους μέσα στο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της... Ε, του Στρασβούργου. Πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα αυτό να είναι συνεναγόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια αυτό είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο υπάρχει με στιγμή στα δικαιωμα το δικαίωμα παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ πρόκειται να εξασφαλίσει κανείς ότι η αγωγή, η προσφυγή θα στρέφεται και κατά των κρατών μελών και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Και ο συνεναγόμενος είναι φυσικά διάδικος πια και εφαρμόζεται σε αυτούς και η απόφαση του δικαστηρίου και έχουν την υποχρέωση να αποδεχθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από μία απόφαση. Δεν είναι απλώς λοιπόν παριστάμενοι στο δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη προσχώρησης θα πρέπει να αναφερθεί αυτή η ιδιαιτερότητα και θα πρέπει να υπάρξει το δικαίωμα αυτό του να παρίσταται η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την ειδικότητα της, του συνεναγόμενου. Έρχομαι τώρα στα, στη δεύτερο ερώτημα για προσφυγές μεταξύ κρατών μελών και θα περάσω στα αγγλικά γιατί στα αγγλικά διατυπώθηκε το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχο το ερώτημα του κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει απόλυτος αποκλεισμό προσφυγών μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν μπορούμε να αναλάβουμε τον κίνδυνο να καθορίσουμε ότι μόνο οι προσφυγές μεταξύ κρατών που εμπίπτουν στον τομέα εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να αποκλείονται. Η δική μου άποψη, αν κατανοώ καλά το ερώτημα, το πρόβλημα που έθεσε ο Ζαν Πολ Ζακέ είναι ότι τότε το ΕΔΑ θα πρέπει να αποφασίζει τι εμπίπτει ή δεν εμπίπτει στη σφαίρα εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, λεπτό, ακόμα και προβληματικό. Μπορούμε να αποφασίσουμε να εξαιρέσουμε πλήρω τι διακρατικού χαρακτήρα προσφυγέ μεταξύ κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να καταγραφεί στην συνθήκη προσχώρησης γιατί βάσει του άρθρου 34 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό είναι μια υποχρέωση η οποία είναι δεσμευτική στα κράτη-μέλη να μην έχουν, θα πρέπει να απόσχουν από μάλλον, Συγγνώμη, να απόσχουν από το να ζητήσουν από ένα εξωτερικό διαιτητή ή δικαστή να ε, αποφασίσει για θέματα τα οποία άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου. Υπάρχουν λοιπόν οι επιλογες αλλά η περίπτωση τη ιλλανδιας εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου του 1978 είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει, που αναφέρθηκε. Τρίτο θέμα ετέθη το ερώτημα σε σχέση με τη δυνατότητα οι πολίτες τρίτων χωρών να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά ενδεχομένως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρους που εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, δεδομένου του ότι η νομολογία του ΕΔΑΔ ορθά, κατά την άποψή μου, είναι όλο και περισσότερο ανήσυχη σε σχέση με διακριτική μεταχείριση που απορρέει μονάχα από την υπηκότητα ενός διαδίκου, κάτι το οποίο είναι όλο και πιο δύσκολο να το δικαιολογήσει κανείς σε μια δημοκρατική κοινωνία. Για μένα η διαφορά μεταχείρισης που οφείλεται στην υπηκότητα ενός διαδίκου και η διαφορά μεταχείρισης μεταξύ των υπηκών τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία πλευρά και των υπηκών τρίτων χωρών από την άλλη πλευρά, όλο αυτό πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή, γιατί οποιαδήποτε ε, διακριτική μεταχείριση δεν είναι κατά διά, διάκριση. Αυτό μπορεί να ισχύει, παραδείγματος για τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά υπάρχουν άλλα θέματα, όπω τα θέματα διαμονή. Δικαιώματο διαμονής και δικαιώματο Ελεύθερη κυκλοφορίας που απαιτούν μια, μια προσεκτική εξέταση. Και αυτό με φέρνει στο τέταρτο ερώτημα που έχει να κάνει με τις ενδεχόμενες επιφυλάξεις που μπορεί να διατυπωθούν, να διατυπωθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την προσχώρησή της στην ΣΥΓΜΑ Είναι το ερώτημα του κυρίου Μέντες Δεβίγα. Υπάρχουν δύο επιφυλάξει που ίσω πρέπει να τι εξετάσουμε σε σχέση με τη σκοπιμότητά του. Η πρώτη θα ήταν να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα εσωτερικά ένδικα μέτρα, μέσα τα οποία πρέπει να εξαντληθούν για να μπορέσει να ευδοκιμήσει μία προσφυγή στο ΕΔΑΔ, ότι αυτά τα εσωτερικά ένδικα μέσα δεν θεωρούνται ότι έχουν εξαντληθεί παρά μόνο εάν ο ενάγων έθεσε το θέμα της συμβατότητος με τα θεμελιώδη δικαιώματα που εγγυάται η ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον ενός εθνικού δικαστή, ζητώντας να υπάρξει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αυτός ο καλύτερο τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου θα έχει τη δυνατότητα να εκφέρει γνώμη πριν το ΕΔΑΔ οδηγηθεί να πάρει μια απόφαση και προφανώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου θα αδράξει αυτή την ευκαιρία που του δίδεται για να εξασφαλίσει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια δεύτερη ενδεχόμενη επιφύλαξη που μπορεί να διατυπωθεί αφορά την έννοια της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από μερικά χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρθηκε στην συμβατότητα με το άρθρο 14 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την μεταχείριση, την διαφορετική μεταχείριση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών τρίτων χωρών. Αυτός είναι ένας χώρος αυτός ο οποίος είναι υπό εξέλιξη, αν τώρα, κάτι το οποίο εγώ δεν θα ήθελα γίνεται, να μην υπάρχει έλεγχος του ΕΔΑΔ για το θέμα αυτό, θα μπορούσε να διατυπωθεί μια επιφυλάξη από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως δεν θα με έβρισκε σύμφωνο. Ευχαριστώ. Το λόγο στην κυρία τη Επιτροπή υπεύθυνη για θέματα Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιώματα των πολιτών για να οργανωθούμε καλύτερα. Ήθελα να συζητήσω, κύριε Ρέντινγκ, μπορείτε να μείνετε μέχρι το τέλο του χρόνου που είχε προληφθεί ή έχετε κάποιο λόγο για τον οποίο θα πρέπει να φύγετε. Εμεί είχαμε προβλέψει να μιλήσει ο δικαστής Τίμερμανς πρώτα και μετά εσείς. και σίγουρα οι συνάδελφοι θα έχουν να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Θέλετε να μιλήσετε πρώτοι, πάντως ερωτήσεις θα γίνουν. Δεν έδωσα ακόμη το λόγο στον καθηγητή Έγγελ, θα μπορούσαμε να το δώσουμε μετά στον δόκτωρα Έγγελ. Πρώτον, η Επίτροπος να μας πει πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή της. Επίτροπος. Κύριε Πρόεδρε, όπως φαντάζεστε, στην πολιτική συχνά υπάρχουν υποχρεώσεις απρόβλεπτες. Κανονικό δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ τώρα. Είμαι εδώ. Θα κάνω την παρέμβαση που είχε προβλεφθεί. Έχει έρθει ο Ιωάννης Κρέμερ, ο οποίος είναι υπεύθυνο των νομικών υπηρεσιών, υπεύθυνο για το θέμα αυτό, αρμόδιος για το θέμα αυτό, θα απαντήσει στο όνομα της Κομισιόν στις ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να κάνω την παρέμβασή μου, κυρίως διότι χθες η Κομισιόν αποφάσισε για την διαπραγματευτική εντολή. Να σας πληροφορήσω γι' αυτό, γι' αυτή την εντολή. Πρόεδρος. Μάλιστα. Αν μπορούτε να μας δώσετε λίγα λεπτά χρόνο για διευθυντικές ερωτήσεις μετά την παρέμβασή σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, έχω μαζί μου τον κύριο Χάνε Κρέμερ, ο οποίο είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Αυτό στο όνομα τη Κομισιόν χειρίζεται το θέμα. Είναι ένα θέμα που, είναι, που το χειρίζονται οι νομικές υπηρεσίες τεχνικά. Πολιτικά ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίο εκπροσωπείται από το πρόσωπό μου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, όπως ήδη είπα χθε, ήταν η μέρα που ολοκληρώθηκε η εργασία του Συλλογικού Σώματος των Επιτρόπων σε συνεργασία με τις νομικές υπηρεσίες και συμφωνήσαμε την εντολή για τις διαπραγματεύσεις η οποία δόθηκε στο Συμβούλιο το Συμβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει και αυτό με την εντολή αυτή πριν προχωρήσουμε. Όπως προβλέπετε στους κανόνες, το Κοινοβούλιο πληροφορείται πλήρως για την εντολή αυτή και το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και μπρος. Η προσχώρηση σύμβαση, όπως ξέρετε, ολοκληρώνει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν είναι ένα ναι. νέο θέμα. Θυμάμαι το 1994 το δικαστήριο του Λουξεμβούργου ήδη είχε γνωμοδοτήσει και είχε πει ότι δεν υπάρχει νομική βάση. Η συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί αυτή τη νομική βάση. Η προσχώρηση δεν είναι προαιρετική πράξη, είναι υποχρέωση. Βέβαια, η σύμβαση είναι μία από τις τέσσερις συνιστώσεις μιας συγκεκριμένης πολιτικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα για την Ένωση. Πρώτον έχουμε τη χάρτα, που είναι τμήμα της Εθνικής Λισαβόνας και που εγώ θεωρώ το, το πιο σύγχρονη κωδικοποίηση θεμελιωδών δικαιωμάτων στον κόσμο. Είναι νομικά δεσμευτική για 27 χώρες. Μεγάλο βήμα στην πολιτική μας δέσμευση υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εμπερέχει όλα τα, δικαίωμα, τα δικαιώματα που έχει και η Σύμβαση. Το νόημα και η εμβέλεια αυτών των δικαιωμάτων είναι το ίδιο με αυτόν που ορίζει η Σύμβαση, αλλά η χάρτα πάει πέραν αυτών. Έχει και άλλα δικαιώματα και αρχές, όπως οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που προέρχονται από τις κοινέ συνταγματικέ παραδόσεις των κρατών μελών και από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και έχει και τα θεμελιώδη δικαιώματα τρίτης γενιάς, που είναι κάπως πιο πρωτότυπα προστασία των ατομικών δεδομένων, data, εγγύησης βιοειφικής, ε, χρηστής διακυβέρνησης. Το άρθρο 53 ορίζει ότι το επίπεδο προστασίας της χάρτας θα πρέπει να είναι εξίσου τουλάχιστον όσο και της σύμβασης. Τώρα πάει πέραν του επίπεδου προστασίας της σύμβασης. Δεύτερο νέο στοιχείο η πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως τα προβλέπει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Χθες στην Κομισιόν πιέσαμε για να υπάρξει ένα πρόγραμμα δράσης με βάση το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Κινούμαστε γρήγορα όπως βλέπετε. Αυτό το πρόγραμμα δράσης ορίζει το πενταετή προγράμματα και για την Επίτροπο Μάλστρομ εκ μέρους των ιστορικών υποθέσεων και για την Επίτροπο Ρέντινγκ σε θέματα δικαιοσύνης και δικαιωμάτων. Ελπίζουμε αυτό να εγκριθεί πριν το καλοκαίρι τρίτο στοιχείο συνιστόσα. Ο πρόεδρος της Κομισιόν χώρισε το χαρτοφυλάκιο σε ένα εσωτερικό υποθέσεων και σε ένα χαρτοφυλάκιο δικαιοσύνη. Αυτό δείχνει τη σημασία που αποδίδει στην ενίσχυση αυτού του χώρου δράσης της Κομισιόν. Σωστά, διότι επιτέλου έχουμε τα εργαλεία για το θέμα τμήμα δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα της συνθήκης να μπορούν να προωθηθούν. Ενώ όσο είχαμε τον τρίτο πυλώνα ως βάση για τις αποφάσεις, δεν μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα και δεν έγιναν πολλά πράγματα. Και ό,τι έγινε ήταν κάπως χαοτικό. Και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί πρακτικά γιατί κάτι που δεν, έλειπε κάτι που δεν μπορούσε να αποφασιστεί με διάταγμα. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Βέβαια, η προσχώρηση στη σύμβαση είναι μια πράξη πολιτική και νομική ιδιαίτερα σημαντική. Από τη σκοπιά των πολιτών θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δίνεται μια εγγύηση σε οποιοδήποτε θεωρεί τον εαυτό του θύμα παραβίαση των θεμελιών δημάτων από ένα θεσμικό όργανο, από ένα όργανο τη Ένωση. και μπορεί να προσφύγει κατά της Ένωσης στο Στρασβούργο κατά του ίδιου όρου, όπως αυτό που ισχύει για προσφυγές κατά των κρατών μελών. Πρέπει να είναι σαφές για τους πολίτες. Πρέπει πρώτα να εξαντληθούν νομικές ό,τι νομικές δυνατότητες, εθνικές δυνατότητες υπάρχουν πριν προσφύγουν σε αυτό το δικαστήριο. Πολιτικά προσχώρηση σημαίνει ότι η Ένωση επιβεβαιώνει και πάλι τον ε, σημαντικό ρόλο για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της στην Ένωση πέραν των συνόρων των 27. Και είναι σημαντικό αυτό. Διότι προσυπογράφοντας την σύμβαση, προσχωρώντας τη σύμβαση, ενισχύουμε το σύστημα του Στρασβούργου εξωτερικού δικαστηριακού ελέγχου για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενοποιώντας τη νομική τάξη των συστημάτων ελέγχου και έτσι ενισχύοντας την αξιοπιστία και εσωτερικά και εξωτερικά της δέσμευσης της Ένωσης υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομικά δε πρώτον συμπληρώνουμε την εισαγωγή ενός νομικά δεσμευτικού χάρτη θα φροντίσουμε η νομολογία και των δύο δικαστηρίων Λουξεμβούργου, Στρασβούργο να εξελίσσεται παράλληλα και είναι μια ευκαιρία να έχουμε ένα σύστημα που να μην έχει ανακολουθίες όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλη την Ήπειρο με υπόσχεση ότι η Ευρώπη όντως θα είναι ενωμένη και με τον νόμο και με τις αξίες. Έπειτα η προσχώρηση δίνει τη δυνατότητα πράξεις που έχουν εγκριθεί από όργανα της Ένωσης άμεσα να αποδίδονται στην Ένωση αντί να αποδίδονται ή άμεσα ή έμεσα σε 27 χώρες, ατομικά ή συλλογικά. Δηλαδή η διομορφία της Ένωσης ως χωριστή νομική ονότητα με αυτόνομες εξουσίες θα αντικατοπτρίζεται αντίστοιχα και επαρκώς στις, ε, στη διαδικασία στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Έπειτα η Ένωση έχει στη διάθεσή της όλα τα δικαιώματα που δίνει η Σύμβαση στους ε, διάδικους προκειμένου να ε, προσπίσουν τα διάφορα δικαιώματα τα οποία θα φτάνουν μέχρι το Στρασβούργο και θα εκπροσωπείται με έναν Ευρωπαίο δικαστή στο δικαστήριο. Το πρωτόκολλο Τη συνθήκη της Λισαβόνας απαιτεί ουσιαστικές εγγυήσεις για μια συμφωνία για την προσχώρηση έτσι ώστε τα ειδικά χαρακτηριστικά του, του νομοθεσίας της Ένωσης να προστατεύονται. Δηλαδή, η εντολή που είναι σύσταση στο Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη αυτού του ε, Υπάρχει αυτό και στην έκθεση της ε, εισηγήτριάς σας. Πρώτον, είναι σαφές ότι οι αρμοδιότητες της Ένωση και οι εξουσίες των οργάνων, όπως ορίζει η συνθήκη, δεν θα επηρεάζονται από την προσχώρηση. Ένας όρος στη συμφωνία προσχώρησης το επιβεβαιώνει αυτό. Επίσης, η προσχώρηση της Ένωσης δεν θα επηρεάσει ούτε την κατάσταση των επιμέρους κρατών μελών σε σχέση με την ΕΣΔΑ ως προς ή τα πρωτόκολλα ή τις επιφυλάξεις. Οι διαπραγματεύσει θα φροντίσουν έτσι ώστε η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει υποχρεώσεις μόνο σε σχέση με πράξεις και μέτρα που έχουν εγκριθεί από τα πρωτοκολλα η τις επιφυλαξεις οι διαπραγματευσεις θα φροντισουν ετσι ωστε η συμφωνια αυτη θα δημιουργησει υποχρεωσεις μονο σε σχεση με πραξεις και μετρα που εχουν εγκριθει απο τα οργανα της Ένωσης όργανοι ή της Ένωσης. Δεύτερον, γιατί προσχώρησε στη σύμβαση που αναφέρεται στο σχέδιο έκθεση της εισηγήτριά σας. Τέσσερα από τα πρωτόκολλα δεν έχουν επικυρωθεί από όλες τις χώρες μέλη. Και ως θέμα πολιτική δαθμιολιά δικαιώματα η Κομισιόν θεωρεί ότι οποιοδήποτε από τα πρωτόκολλα αυτά μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την άσκηση των εξουσιών της Ένωσης. Ορισμένες εγγυήσεις που υπάρχουν στα πρωτόκολλα αυτά αντικατοπτρίζονται στη χάρτα. Μία προσχώρηση λοιπόν της Ένωσης στα πρωτόκολλα αυτά είναι άκρος επιθυμητέα ως θεμαρχής. Ωστόσο αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, τα κράτη-μέλη ακόμα είναι διαρρημένα στο θέμα της προσχώρησης της Ένωσης στα συγκεκριμένα αυτά πρωτόκολλα που δεν έχουν επικυρωθεί από όλες τις χώρες. Συνεπώς η Κομισιόν προτείνει μια μέθοδο δύο χρόνων προκειμένου να υπάρξει μια, ε, μια ε, συμφωνία για τη διαπραγματευτική εντολή. Η πρώτη φάση, δικαίωμα πρόσβασης προσχώρησης σε οποιοδήποτε από τα πρωτόκολλα της σύμβασης, δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης και δεύτερη φάση μετά να αποφασίσουμε σε ποια πρωτόκολλα θα προσχωρήσουμε πέραν της σύμβασης της ίδιας. Θέλουμε να γίνει ομαλή ένταξη της Ένωσης στο σύστημα της σύμβασης. Αυτή η προσχώρηση λοιπόν θα πρέπει να προστατεύσει τα ουσιαστικά διαδικαστικά χαρακτηριστικά του συστήματος. Πρέπει να πληρούνται δύο κριτήρια. Πρώτον, τα ειδικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας της Ένωσης πρέπει να προφυλαχθεί και δεύτερον έχουμε τις ειδικέ καταστάσεις της Ένωσης ως χωριστής νομικής προσωπικότητας με αυτόνομες εξουσίες που θα είναι ε, διάδικο με, μέλος παράλληλα με τα κράτη-μέλη με ένα συγκεκριμένο μηχανισμό που ουσιαστικά έχει οριστεί για κράτη μόνον με τεχνικές και διαδικαστικές τροπολογίες της σύμβασης που απαιτούνται προκειμένου να πληρούνται αυτά τα δύο κριτήρια, θα ήθελα να αναφέρω το μηχανισμό του co-defendant, αυτού του συνεναγόμενου που πρότεινε χθε η Κομισιόν. Χαίρομαι για το ότι ο μηχανισμός αυτός του συνεναγόμενου ε, συνιστάται και στο σχέδιο έκθεσης του Κοινοβουλίου. Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο η Ένωση να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ως συνεναγόμενος στις διαδικασίες όταν έχουν προσφυγεί κατά κράτους μέλους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η υποτιθέμενη παραβίωση της σύμβασης αφορά μία πράξη που το κράτο μέλος ενέκρινε για να συμμορφωθεί με υποχρέωσή του με βάση την νομοθεσία της Ένωσης. Και όταν το κράτο μέλος το συγκεκριμένο θα μπορούσε να το είχε αποφύγει παραβιάζοντας μόνο την ε, νομοθεσία της Ένωσης. Άρα μη τηρώντας τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την νομοθεσία της Ένωσης. Μόνο αν έχει λοιπόν πλήρες καθεστώς ε, συμμετέχοντος στην ε, δικαστηριακή διαδικασία με όλα τα δικαιώματα που αυτό σημαίνει προκειμένου, για την Ένωση προκειμένου να προστατεύσει την θέματα κοινωτική νομοθεσίας και της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και την, ε, το δικαίωμα να γίνει προσφυγή στο ανώτατο σώμα του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, έτσι, η Ένωση θα, είναι, θα δεσμεύεται εξίσου αποφάσεις από το Δικαστήριο του Στρασβούργου αν υπάρχει παραβίαση της σύμβασης και θα είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει την απόφαση αυτή του Δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση μπορεί να είναι υποχρεωμένη να καταργήσει, ή να τροποποιήσει ένα τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης. Αν δεν είχαμε αυτό το μηχανισμό του συνεναγόμενου, το, το δικαστήριο του Στρασβούργου θα μπορούσε να πάρει μια απόφαση μόνο κατά μιας χώρας μένος, ακόμα και αν η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, προερχόταν από νομοθεσία της Ένωσης. Οπότε το κράτος μένος δεν θα μπορούσε να εκτελέσει μια τέτοια εντολή. Δεν μπορεί να καταργήσει, να τροπολογήσει ε, τη συγκεκριμένη νομοθεσία της Ένωσης, θεωρούμε ότι το, Δικαστήριο του Στρασβούργου καταρχήν δεν θα πρέπει να ερμηνεύει νομοθε... την νομοθεσία της Ένωσης. Γιατί η αρχή της αυτόνομης ερμηνείας του νόμου που το έχει η Ένωση, θα λόγω αυτού θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά κράτος μέλος και όχι μόνο σε περιπτώσεις που η πράξη που υποτίθεται παραβιάζει την σύμβαση καθορίζεται μόνο από νομοθεσία της Ένωσης. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιεί εσωτερικούς κανόνες για να ορίσει ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε η Ένωση να παίρνει μέρος στην διαδικασία ως συνεναγόμενος. Η εισαγωγή λοιπόν του μηχανισμού κόντι φέναν συνεναγόμενο είναι μια μικρή αλλαγή στην σύμβαση. Είναι τεχνική, είναι διαδικαστική και δεν στρεβλώνει την σωστή λειτουργία της σύμβασης της Το αντίθετο εξασφαλίζει μια ομαλή ένταξη της Ένωσης στο σύστημα της σύμβασης. Θεσμικά δε, η θέση της Κομισιόν είναι ότι οι εκπρόσωποι της Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχουν στα όργανα της Σύμβασης σε ίση βάση με εκπροσώπους άλλων συμβολωμένων μερών. Κυρίως αυτό αφορά το δικαστήριο του Στρασβούργου. Η παρουσία ενός δικαστή που θα έχει εκλεγεί από κάθε συμβολώμενο μέρος είναι μια από τις βασικές αρχές της συνθήκης. Είναι μια αρχή που μας εξασφαλίζει ότι κάθε νομικό σύστημα θα εκπροσωπείται στο δικαστήριο και αντικατοπίζει και τη σύστημα συλλογική εγγύησης που προβλέπεται από τη Σύμβαση για κάθε συμβαλόμενο μέρος με, συμμετοχή, με συμμετέχοντες και ενισχύει την νομιμότητα των αποφάσεων που παίρνει το δικαστήριο. Άρα η αρχή της παρουσίας ενός δικαστή που έχει εκλεγεί από την Ένωση είναι ένα must. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης επειδή το δίκαιο της Ένωσης είναι αυτόνομο, ειδικό και ένα από τα κύρια ωφέλη αυτής της προσχώρησης είναι το ότι το νομικό σύστημα της Ένωσης εκπροσωπείται επαρκώς και στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο έχει την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται και να λάβει υπόψη τις ιδιομορφίες του δικαίου της Ένωσης. Η Κομισιόν λοιπόν είναι υπέρ του να υπάρχει ένας μόνιμος δικαστής, πλήρες μέλος, που να έχει εκλεγεί από την Ένωση με το ίδιο καθεστώς, με, τα, με τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως και οι άλλοι δικαστές, και που να παρεμβαίνει ενδεχομένω σε όλες, να μπορεί να παρεμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Η μέθοδος εκλογής του δικαστή. Και στρέφομαι τώρα στο Κοινοβούλιο συνήθις διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση θα πρέπει να ισχύει αυτό σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική συνδιάσκεψη επιλέγει ένα δικαστή βάσει ενός καταλόγου τριών υποψηφίων που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ, αυτό είναι κοινοβουλευτικό ζήτημα βέβαια, θεωρώ ότι ένας ε, κατάλληλος αριθμός, ένας επαρκής αριθμός μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ε, αυτή συνέλευση όταν εκλέγει αυτή τους δικαστές του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Η θέση της Κομισιόν και πάλι συνάδει με τα όσα λέγονται στο σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, χαίρομαι πολύ που ένα τέτοιο επικοδομητικό πνεύμα συνεργασίας υπάρχει με την Ισπανική Προεδρία. Η Ισπανική Προεδρία έδειξε μεγάλη προθυμία στην εκπόνηση της εντολής. Έχει κατατεθεί τώρα στο Συμβούλιο και ελπίζω ότι το Συμβούλιο πολύ γρήγορα θα εργαστεί επί της εντολής αυτής έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τις προσχωρήσεις το συντομότερο δυνατόν. Πρόεδρε. Θα καταλάβατε ότι η Κομισιόν δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην εντολή αυτή και με πολύ μεγάλη σοβαρότητα θα διαπραγματεύσεις και η Κομισιόν να σας πω ότι διαπραγματεύεται και εν το χρόνο θα ενημερώσει το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία και σε συνεχή συνεργασία με το δικαστήριο και με τους συμβούλους που μπορούν να μας βοηθήσουν προκειμένου να ολοκληρωθούν ταχαίως οι διαπραγματεύσεις, γιατί όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει και όλη τη διαδικασία, γιατί τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της κύρωσης. Και να σας πω ότι ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με τους 27, αλλά υπάρχουν και 20 ακόμα μέλη και μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος. Ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο. Να σας ρωτήσω αν είναι δυνατό τα μέλη της Επιτροπής να δουν το σχέδιο κειμένου για την εντολή. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Τώρα εσείς πρέπει να φύγετε. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να σας υποχρεώσουμε να μείνετε εδώ με τη βία. Σας ευχαριστώ. Πάντως πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε με την Κομισιόν πολύ στενά για τα ζητήματα αυτά.

Λυπούμαστε που δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε σε ανάκριση την Επιτροπό μας, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε και αλλιώς ε, την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της εδώ. Τώρα, σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο, είχαμε μείνει στο εξή. Θα έπρεπε να ακούσουμε την ενδεχομένη απάντηση του κυρίου Έγγελ. Δεν ξέρω, μήπως ε, θα ήταν καλύτερο να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στο δικαστή Τίμερμανς από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν στο πλαίσιο της συμπληρωματικής συζήτησης θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τον κύριο Έγγελ. Παρακαλώ λοιπόν ε, το δικαστή Τίμερμαν να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ καταρχήν που καλέσατε ένα μέλος του δικαστηρίου να παραβρεθεί στην ακρόαση αυτή. Είναι προφανές ότι εδώ δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος του δικαστηρίου. Το δικαστήριο δεν έχει επίσημη θέση για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα. Όμως ε, τα μέλη του δικαστηρίου σκέφτονται φυσικά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όπως και να έχει θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι εγώ θα τοποθετηθώ προσωπικά. Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για την ερώτηση που τέθηκε επανειλημμένω. Ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία τη προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΣΔΑ. Δεν πιστεύω προσωπικά ότι το επίπεδο προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, όπως διασφαλίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Χάρτα και από την ομολογία τη Ένωση, ε, δεν είναι ικανοποιητικό και ότι η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ θα είναι απαραίτητη για να καλυφθούν κάποια κενά. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη εφαρμόζει τη σύμβαση όπως γνωρίζετε στην ομολογία του. Τα τελευταία χρόνια αναφέρεται σε θέματα αυτά όλα ένα και λεπτομερέστερα. Όλο ένα και λεπτομερέστερα αναφέρεται λοιπόν στην ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και μάλιστα και άτυπα να σας πω ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο δικαστηρίων είναι εξαιρετική. Μπορώ να το πω αυτό, σχεδόν είμαι μέλος πλέον του δικαστηρίου. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Υπόθηκε ήδη, αλλά θέλω να το τονίσω κι εγώ. Η θέση σε ισχύ τη συνθήκη στη Λισαβόνα. Από τη στιγμή τη θέση σε ισχύ έγινε δεσμευτική η ΕΣΔΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δυνάμει και της χάρτας. Έχουμε το άρθρο 52 παράγραφος 3 της χάρτας που μας λέει ότι όταν ε, τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη χάρτα αποκρίνονται σε δικαιώματα που υπάρχουν στη σύμβαση, τότε είναι το πεδίο, το βεληνικές τους είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε σύμπτωση ε, τέτοια των δικαιωμάτων, θα πρέπει να έχουμε την ελάχιστη προστασία. Δηλαδή, ήδη σεβόμαστε τη σύμβαση, αλλά και την ομολογία ε, του Δικαστηρίου του Στρασβουργού. Αυτό επιβάλλεται στην Ένωση. Πρόκειται για μια υποχρέωση σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου. Αν ε, έτσι έχουν τα πράγματα, ε, δηλαδή η σύμβαση είναι ήδη ευρέως δεσμευτική για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να προσχωρήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο προφανείς λόγοι. Καταρχήν, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενταχθεί στο πανευρωπαϊκό σύστημα της εγγύησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι όπως δυσφαλίζονται από, από την ΕΣΔΑ και το ΕΔΑΔ, και ο δεύτερος λόγος ε, είναι ότι όλοι ε, γνωρίζουμε ότι όταν ε, υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τότε θα πρέπει να υπάρχει προσφυγή κατά των κρατών μελών, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Αυτά σχετικά με την προστιθέμενη αξία. Η προσχώρηση λοιπόν είναι σκόπιμη και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της συνθήκης είναι απαραίτητη. Όμως ε, η υλοποίηση της θα επιφέρει κάποια προβλήματα που συζητήσαμε σήμερα και το πρωί και μάλιστα ορισμένα προβλήματα είναι αρκετά πολύπλοκα και προκαλούνται από την ιδιαιτερότητα του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρωτόκολλο υπερθυμών 8 ε, ότι οι υπογράφοι Συνδίκη Λισαβόνας γνώριζαν ε, ότι η προσχώρηση θα πρέπει να σεβαστεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου της. Και μάλιστα δεν θίγονται οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε των οργάνων της. Θα ήθελα τώρα να τονίσω πιο συγκεκριμένα ένα από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ένωσης. Πρόκειται για μια επιπλοκή που προκύπτει από το ότι, ένας, ότι γενικά η δράση της Ένωσης έχει συνέπειες για τους πολίτες μέσω εθνικών μέτρων εφαρμογής. Ακόμη και αν υπάρχουν ε, κανονισμοί οι ε, οποίοι δεν άπτονται στην εφαρμογή εθνικών μέτρων, αλλά εφαρμόζονται απευθείας. Ε, μόνο κατά εξαίρεση οι πολίτες, οι ιδιώτες μπορούν απευθείας να προσφύγουν κατά τον κανονισμών αυτών σε δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης. Για να υπάρξει προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι πολίτες κανονικά θα πρέπει να προσφύγουν ε, στα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα και τελικά στις εθνικές δικαιοδοσίες, στα εθνικά δικαστήρια και αν ε, σε κάποια περίπτωση δεν υπάρχει επαρκής προστασία από τον εθνικό δικαστή, τότε οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν ε, στο δικαστήριο του Στρασβούργου αφού θα έχουν εξαντληθεί τα εθνικά ενδικά μέσα. Πράττοντας αυτό, οι πολίτες μέσα μπορούν να αμφισβητήσουν τη δράση της ε, Ένωση ε, που τίθεται σε εφαρμογή από τα εθνικά μέτρα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο ιδιώτη σήμερα, ο πολίτη, πριν από την προσχώρηση, δεν σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα τελικά να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου, αλλά η δυνατότητα αυτή υπάρχει μόνο... Ε, όταν προσφεύγει κατά των κρατών μελών. Όταν θα έχει προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να καταδικαστεί από το Δικαστήριο του Στρασβούργου όταν είτε έμεσα ή έμεσα μία δράση της Ένωσης αμφισβητείται. Και φυσικά η συμφωνία της ενωσης αμφισβητειται και φυσικα η συμφωνια τη προσχώρηση θα πρέπει να ρυθμίζει και τη συμμετοχή τη Ένωση σε αυτή, τη διαδικασία. Το συζητήσαμε λεπτομερό σήμερα το πρωί. Όμως εδώ έχουμε μια σοβαρή δυσκολία ενώπιόν μας πρόκειται για την ευθύνη και την κύρια λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου να διασφαλίσει το σεβασμό του δικαίου της Ένωσης και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και όταν το πρωτόκολλο 8 απαιτεί προσχώρηση στη σύμβαση να γίνει υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων ε, των κοινοτικών οργάνων. Αυτό σημαίνει, στοχεύει και στην αρμοδιότητα στην ευθύνη του δικαστηρίου. Έτσι λοιπόν, σε όλες σας περιέγραψα, Υπάρχει μόνο μία δυνατότητα το δικαστήριο να λάβει αυτή την ευθύνη με την προδικαστική διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα και εν τέλει την υποχρέωση τα εθνικά δικαστήρια να στείλουν προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν ε, τελικά η δράση της Ένωσης ε, συνάδει, σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όμως ε, ο ιδιώτης δεν έχει αυτή την πρόσβαση να υποβάλει το δικαστικό ερώτημα, το αποφασίζει αυτό ο Εθνικός Δικαστής. Ο πολίτης μπορεί να ζητήσει από το δικαστή να χρησιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία, να θέσει προδικαστικά ερωτήματα, αλλά δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει. Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με όσα υπόθηκαν από τον ε, κύριο Ζακέ σήμερα το πρωί, εγώ προσωπικά νομίζω ότι εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί, Γιατί θεωρώ ότι είναι δύσκολο αποδεκτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή μάλλον το Δικαστήριο του Στρασβούρου διορθώνει ο μιλητή, να μπορεί να καταδικάσει την Ένωση για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, αν το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου δεν είχε πρώτο τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα αυτό. Και μάλιστα αναρωτιέμαι αν μια τέτοια συνέπεια δεν θα αντίκειτο στην αρχή της εξάντλησης των ένδικων μέσων, έτσι όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στο ψήφισμα, στην απόφαση του δικαστηρίου 3 Σεπτεμβρίου 2008 στην ε, υπόθεση Κάντι. Είχαμε εκεί δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, μια υπόθεση τρομοκρατίας, ε, όπου το δικαστήριο καθόρισε τις αρχές βάσει των οποίων όλες τις κοινωνικές πράξεις θα πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραθέτω το δικαστήριο πρέπει να ελέγξει ε, αν ε, έχει γίνει σεβαστό το σύστημα της ε, προσφυγής των ένδικων μέσων όπως προβλέπεται στις συνθήκες. Έτσι λοιπόν πρέπει να προβλεφθούν όπως και να έχει μηχανισμοί που επιτρέπουν στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου να τοποθετηθεί μια υπόθεση πριν να αποφασίσει, πριν να τοποθετηθεί το δικαστήριο του Στραμβούργου. Ποιο μηχανισμό. Μια πρώτη επιλογή θα μπορούσε να είναι να καθορίσουμε την εξάντληση των ένδικων μέσων στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή ε, μία προσφυγή στο δικαστήριο του Στρασβούργου να είναι δυνατή αφού το δικαστήριο του Λουξεμβούργου θα έχει μπορέσει να τοποθετηθεί με προδικαστικό ερώτημα. Βέβαια, όταν ε, η Εθνική Δικαιοδοσία έχει στείλει αυτό το προδικαστικό ερώτημα στο Λουξεμβούργο, θα πρέπει να περιμένουμε την έκθεση της προδικαστικής διαδικασίας και της εθνικής διαδικασίας, Είναι προφανέ. Όμως, αν δεν υπάρχει αυτή η προδικαστική διαδικασία, το να αποκλείσουμε ε, την ε, πρόσβαση στο δικαστήριο του Σουρβούργου δεν φαίνεται ικανοποιητική γιατί πρέπει να προστατεύονται τα δικαιώματα του ιδιώτη και του πολίτη κυρίως γιατί αυτός ο πολίτης δεν ελέγχει την πρόσβαση στην προδικαστική διαδικασία δεν μπορεί να ελέγξει κατά κανένα τρόπο τη χρήση της διαδικασίας αυτής και το να απαιτείται ως απέτηση του παραδεκτού ε, μιας προσφυγής στο δικαστήριο του Στρασβούργου να έχει εξαντληθεί ε, η προσφυγή στην προδικαστική διαδικασία δεν φαίνεται να είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό για λόγους αρχής αλλά μάλλον για λόγους πρακτικούς. εμείς θα πρέπει να δούμε, δεν θα είναι μάλιστα ιδιαίτερα σκόπιμο να ε, απαγορεύσουμε να υπάρχει αυτό το πέρασμα από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Η πρώτη δηλαδή εναλλακτική δεν φαίνεται λογιστική. Δεύτερη τώρα εναλλακτική το δικαστήριο του Στρασβούργου θα μπορούσε να θεωρήσει απαράδεκτη μία προσφυγή σε ένα πλαίσιο που θεωρεί ότι ο εθνικός δικαστής θα έπρεπε να έχει στείλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αναφέρω αυτή την εναλλακτική γιατί την έχουμε ήδη στην ομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Υπάρχει μια ομολογία σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο του Στρασβούργου επαλήθευσε αν η απουσία προδικαστικού ερωτήματος είναι αυθαίρετη ή όχι και επομένως αντίκειται ε, στο δικαίωμα της δίκαιης δίκης που δικαιούται το άρθρο 6 της Σύμβασης. Όμως ε, το ίδιο το θέμα του αυθαίρετου σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ιδιαίτερα εξαιρετικές καταστάσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υποχρέωση των ε, εθνικών δικαστηρίων ε, να ε, προσφύγουν στην προδικαστική διαδικασία δεν είναι κάτι απόλυτο. Υπάρχει αναγκαιότητα να απαντηθεί καταρχήν το θέμα, δηλαδή να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τη διένεξη σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, είναι σημαντικό να δούμε αν το δικαστήριο του Στρασβουργού θα ε, έχει ένα πιο αυστηρό έλεγχο. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα, γιατί τελικά το λόγο δικαστήριο θα ασκήσει την αυτόνομη θα την αυτόνομη αρμοδιότητα που έχει το Εθνικό Δικαστήριο να στείλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και επίσης το Δικαστήριο του Στρασβούργου ε, ουσιαστικά θα έρθει εδώ να επισέλθει σε ένα θεμελιώδη ζήτημα που έχει να κάνει με την προδικαστική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα το πρωί αναφέρθηκε ότι ο ενάγων τουλάχιστον θα πρέπει να προτείνει στον εθνικό δικαστή να εφαρμοστεί η προδικαστική διαδικασία, αλλιώς θα πρέπει να θεωρείται μη παραδεκτή η προσφυγή του ενώπιον του ΕΔΑ, διότι δεν υπήρξε εξάντληση των ενδικών μέτρων, μέσων. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια επαρκή απάντηση στο πραγματικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Αλλά λόγω ελλείψεως χρόνου δεν θα μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειε, γιατί ήθελα να προτείνω και μια τρίτη ε, πρόταση, μια τρίτη λύση στα λίγα λεφτά που μου μένουν. Για μένα θα ήταν προτιμότερο να προβλέψουμε ένα μηχανισμό, όχι μονάχα σε επίπεδο του Δικαστήριου του Στρασβούργου, του ΕΔΑΔ, <clears throat> αλλά καταρχήν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε, παραδείγματο χάρη, να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από το Δικαστήριο του Λουξεμβούρου να εκφέρει άποψη σε σχέση με το συμβατό μιας πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ακόμα αν πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με, ένα, με την περίπτωση που μία προσφυγή έχει θεωρηθεί ότι δεν ήταν παραδεκτή από το δικαστήριο του Στρασβού. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι συμμετέχον σε μια τέτοια διαδικασία σε αυτή την περίπτωση και τότε θα υπάρχει δυνατότητα να εκτιμήσει το σκόπιμο του να υπάρξει μια αίτηση στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου για το κατά πόσον θα έπρεπε να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Στρασβούργο. Εάν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα έπρεπε να αναστέλλεται η διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑΤ μέχρι ότου εκδοθεί μια απόφαση από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Εάν αποφασίσει το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου ότι πράγματι υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τότε θα πρέπει να περατωθεί η διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑΔ. Αντίθετα, θα μπορούσε να συνεχιστεί η διαδικασία. Στην μια πρώτη περίπτωση θα διακοπεί, στη δεύτερη θα συνεχιστεί. Και κλείνοντα, κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εγώ να τονίσω ότι με αυτά τα λίγα που είπα ήθελα να σας ευαισθητοποιήσω σε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για, το, για την οποία προσχώρηση είναι απαραίτητο να επιλύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν πριν από την προσχώρηση. Ευχαριστούμε. Ξαναείδαμε πάλι πόσο περίπλοκο είναι τα θέματα. Πάντως μας βοηθάτε να ξεκαθαρίζετε η κατάσταση. Τώρα, στη συζήτηση από εδώ και, ε, που αρχίζει, θα δώσω το λόγο καταρχήν στον δόκτωρα Έγγελ ε, να κάνει μερικά σχόλια από θέματα που μείνανε εκκριμή από το προηγούμενο τμήμα της συζήτησης. Ευχαριστώ. Ένας βουλευτής μου έθεσε ένα ερώτημα που είχε να κάνει με χρήματα, με προϋπολογισμούς, με συμβολή του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσα να απαντήσω σε δύο βήματα, σε δύο στάδια το ερώτημα αυτό. Καταρχήν σε επίπεδο αρχών και μετά σε συγκεκριμένο επίπεδο. Σε επίπεδο αρχών, όταν πρόκειται για την περίπτωση αυτή, δεν είναι μία κατά κάποιο τρόπο πράξη συμφώνου όπου πρέπει να φέρει την πρίκα η νύφη στο γάμο. Εδώ πρόκειται για μια συμφωνία δύο ισοτήμων εταίρων για μια σύμβαση η οποία βασίζεται σε ένα σύνολο αρχών. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα χρήματα τα οποία έχει πάρει από τα κράτη-μελών. Βέβαια, ο προπολογισμό του Συμβουλίου τη Ευρώπη είναι πολύ μικρότερο από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, λοιπόν, πιστεύω ότι μέσα από την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αλλάξει και η αντιμετώπιση ορισμένων Υπουργείων Εξωτερικών. Τα χρήματα τα οποία δίνονται λοιπόν στο ΕΔΑΔ από το Συμβούλιο της Ευρώπης έχουν και μια πολιτική σοδιά, εάν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά με, μαζί τους. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο βάρος εργασίας που έχει να αντιμετωπίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΕΔΑΤ. Αυτό οφείλεται στην διεύρυνση προς τα, ανατολικά του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία είναι παράλληλη με αυτήν την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά. Μετά από την πτώση του κομμουνιστικού στρατοπέδου, είδανε πολύ και εγώ με μεγάλη χαρά ότι υπήρξε υποχρέωση ορισμένων να αποδεχτούν την ύπαρξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη εφαρμογής τους τα μετακομμουνιστικά κράτη θέλησε το Συμβούλιο της Ευρώπης το ταχύτερο δυνατόν να τα συμπεριλάβει, αλλά δεν υπήρχαν ακόμα μέσα στα κράτη αυτά οι απαραίτητες δομές για να αντιμετωπιστούν στο εσωτερικό τους τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξε μια σειρά κρατών στα οποία, για τα οποία οι μισές περίπου διαδικασίες οι οποίες έρχονται στο Στρασβούργο προέρχονται από το γεγονός ότι το αντίστοιχο κράτος δεν εφήρμοζε αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων. Βλέπετε λοιπόν πόσο ασθενείς είναι αυτές οι δομές που υπήρχαν στα κράτη με αυτά τα οποία προσχώρησαν στο Συμβουλίο της Ευρώπης και ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν να καλυφθεί το έλλειμμα των δημοκρατικών ε, δομών στα κράτη αυτά με τον τρόπο αυτό. Εάν τα κράτη-μέλη αυτά ήταν υποχρεωμένα του Συμβουλίου της Ευρώπης να υπογράψουν τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να αναγνωρίσουν την δοσηδικία του ΕΔΑΔ, αυτός θα ήταν ένας μοχλός πίεσης για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη αυτά να κάνουν μια αλλαγή στο εσωτερικό του ένωμο σύστημα για να μπορέσουν να πλησιάσουν το σύστημα του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Αυτό οδήγησε σε μια έκρηξη και πολλαπλασιασμό των προσφυγών ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβού. Σε γενικό επίπεδο τώρα, ο προπολογισμό του ΕΔΑΔ είναι μονάχα ένα μικρό κομμάτι του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και επίσης είναι ένα μικρό τμήμα του προϋπολογισμού του δικαστηρίου για την πρώην Ιουκοσλαβία ή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δηλαδή η... είναι η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ΕΔΑΔ είναι πιο φτηνή μέσα στα εισαγωγικά αυτά σε ό,τι αφορά τα άλλα δικαστήρια. Έχουμε τώρα σε πιο προσωπικές παρατηρήσεις, σε πιο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Αν έχει το δικαστήριο μία αυτονομία σε σχέση με την πρόσληψη και τη διαχείριση του προσωπικού του, και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης πάυσει να αναμειγνύεται στα θέματα προσωπικού του, Ευρωπαϊκού, του Δικαστήριου του ΕΔΑΔ, εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα το οποίο μπορεί να λυθεί άκοπα και χωρίς δαπάνη. Το θέμα της αυτονομίας του προϋπολογισμού του Δικαστηρίου του Στρασβού σημαίνει ότι το Δικαστήριο υποβάλλει μια πρόταση, τι χρειάζεται να έχει και αποφασίζει η Επιτροπή Υπουργών τι θα του δώσει αλλά δεν είναι κάτι που περνάει από το χέρι του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος θα πρέπει να κάνει την πρόταση και την απόφαση για τον προϋπολογισμό του δικαστηρίου, είναι η Επιτροπή Υπουργών, η οποία με διάφανο και ε, εποπτεύσιμο τρόπο θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις αυτές και έτσι το δικαστήριο έχει τη δική του αυτονομία την οποία μπορεί να διατηρήσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι σαφής και διάφανος. Δηλαδή θα ήθελα να κάνω μια έκκληση για μια μεγαλύτερη διαφάνεια και σε ό,τι αφορά το καθεστώς των δικαστών οι κανονισμοί οι οποίοι είναι εμβαλωματικοί και αποσπασματικοί να μπορέσουν να αντικατασταθούν από μια γενική ρύθμιση η οποία περιλαμβάνει συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τους δικαστές του ΕΔΑΤ και αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ομαλοποίησης αυτών των πραγμάτων αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε και αυτό είναι το τελευταίο μου, η τελευταία μου παρα, παρατήρηση ότι για την αποτελεσματικότητα του δικαστηρίου δεν ευθύνονται μόνο οι δικαστέ, αλλά και το προσωπικό υποστήριξη. Δηλαδή οι νομομαθεί που του πλαισιώνουν. Και εδώ εναπόκειται σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη να κάνουν τι απαραίτητε προσαρμογέ. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να πληρώσει χρήματα για να μπει στην δομή αυτή, αλλά αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει τον εαυτό της σαν ένα σύνολο, σαν ένα τμήμα ενό γενικότερου συνόλου στο οποίο έχει κάποιες ευθύνες. Θα πρέπει λοιπόν το πολιτικό σύνολο να αναλάβει τις ευθύνες της απόφασης και επομένως από αυτή την άποψη θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη διεύρυνση της Επιτροπής των Υπουργών για να γίνουν όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λόγω στην συνεισηγήτρια κυρία Γκάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση προς τον δικαστή Τίμερμονς. Σας είμαι ευγνώμων για το ότι αναφέρετε όλους τους μηχανισμούς. Γιατί έτσι μας δείξατε ότι στις λεπτομέρειες αυτές κρύβεται η ουσία. Πώς ένα άτομο δηλαδή, ένας άνθρωπος θα τοποθετηθεί μέσα στο σύστημα αυτό και πώς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε προστιθέμενη αξία για τον κάθε πολίτη. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε. Πρώτον, καταρχήν θα πρέπει να εξηγηθούν όλα τα <clears throat> εσωτερικής φύσεως μέσα Εξαντλώντας αυτά τα εσωτερικά εθνικά μέσα, μπορεί να υπάρχει η ανάγκη για προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού. Δεν υποχρέωσε το Εθνικό Δικαστήριο να το ζητήσει αυτό, αλλά μπορεί να, το, να ζητήσει αυτή την προδικαστική απόφαση το Εθνικό Δικαστήριο. Αλλά ακόμα και αν ζητήσει προδικαστική απόφαση του εθνικού Δικαστήριο, και την πάρει, μετά από πολίτης μπορεί να πάει στο Στρασβούργο. Ήδη έχουν περάσει μίνιμουμ 8 με 10 χρόνια για την ιστορία αυτή. Δηλαδή, για να υπάρχει επιπλέον δυνατότητα, αν το ελάχιστο σε χρόνο είναι μετά από 8 με 10 χρόνια, Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να πείσουμε τον πολίτη ότι είναι προς το καλό του αυτό. Γι' αυτό σας ενθαρρύνω όλους σας δικαστές, εμπειρογνώμονες, εμά, εμάς τους πολιτικούς που είναι η δουλειά μας στην Επιτροπή αυτή εδώ, να προσπαθήσουμε να υπάρξουν μηχανισμοί που θα δίνουν πιο ευέλικτες δυνατότητες κάτι που να είναι πραγματικά προστιθέμενη αξία για τον πολίτη. Αλλιώς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτό είπα στην παρουσίασή μου το πρωί. Μην τυχόν δημιουργήσουμε φρούδες προσδοκίες, υπερβολικές προσδοκίες. Λέμε ότι είναι σημαντικό, είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό και ότι πρέπει να το κάνουμε και ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος δράσης. Αλλά παράλληλα πρέπει να δείξουμε πώς μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο σας συνάδελφο Μέσσερ Σμιτ, σας θυμίζω στο πέρας της πρωινής συνεδρίασης η Επιτροπή μας προσφέρει ε, κάτι που θα μπορείτε να Φάτε έξω από την αίθουσα προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση αν θέλετε. Θα πάει στη διαθήση αυτή η δυνατότητα έξω από την αίθουσα. Μέσα Σμίτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα που ανέφερθηκε πολλές φορές και που είναι κεντρική σημασία. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα θέμα επίδικο μεταξύ της σύμβασης και άλλων κειμένων, το θέμα είναι τι θα ληφθεί ως βάση. Θα πρέπει κανονικά να ληφθεί αυτό που παρέχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια, νομική ασφάλεια. Ποιο είναι το καταλληλότερο δίκαιο στην περίπτωση αυτή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. οι δανέζικε γελιογραφίε για τον προφήτη. Θα μπορούσε κάποιο να πει, ναι, η θρησκευτική ευαισθησία είναι σημαντική. Ένα άλλο όμως μπορεί να πει, η ελευθερία έκφραση είναι πιο σημαντικό και υπερέχει. Άρα το άρθρο 10. Εγώ λέω ότι είναι κάπως υπερβολικό να πάμε ε, στη νομική βάση που δίνει τα περισσότερα δικαιώματα στο ποιος θα κερδίσει χωρίς να δούμε ποιες είναι οι διάφορες συνέπειες αυτής της επιλογής γιατί είναι δύσκολο να κρίνουμε ποιο είναι το καταλληλότερο δίκαιο. Το δίκαιο του προσφεύγοντος ή κάποιο άλλο. Αν έχουμε τη χάρτη από τη μια μεριά και τη σύμβαση από την άλλη, τι θα επιλέξει κανείς. Ερώτημα. Πρόεδρος. Ο δικαστής Τίμερμαν έχει το λόγο για να απαντήσει. Εκτός αν υπάρχει κάποιος άλλος ε, που θέλει να πάρει το λόγο εκ των προτέρων. Πριν. Ίσως θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκάλ. Το κατανοώ και αυτό. Και εγώ εξαρτώμαι από εσά βέβαια για τις απαντήσεις. Ίσως τα αγγλικά. Είδα ότι ήθελα να πάρει το λόγο για κάποιος άλλος από τους εμπειρογνωμονές μας. Και νομίζω ότι ίσως καθώς εσείς ήσασταν αυτός που πήρε το λόγο τελευταίος, καλό θα ήταν να σας δώσουμε κατόπιν το λόγο, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε. Είναι πραγματικά πολύ παθιασμένα τα θέματα που έθιξε ο δικαστής ε, Τίμερμαντς ε, για να διατηρηθεί το μονοπόλιο της ε, ερμηνείας του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να φτιάχνουμε κατασκευάσματα που δεν λειτουργούν για το πολίτη. Εδώ βρισκόμαστε σε κάποιες ε, πολύ σπάνιες ε, περιπτώσεις γιατί το δικαστήριο του Στρασβούργου δεν ερμηνεύει το ε, εθνικό δίκαιο έτσι λοιπόν για την περίπτωση που οι δικαστές του Στρασβούργου θα τρελαίνονταν και θα άρχιζαν να ερμηνεύουν το εθνικό δίκαιο, τότε θα έπρεπε να κατασκευάσουμε κάτι τέτοιο όμως. Κοιτάξτε εδώ, διαφωνούμε, είναι λογικό να ισχύει και κάτι τέτοιο σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως είπε και ο κύριος Δισκούτερ η τεχνικές εξάντλησης των εσωτερικών ένδικων μέσων έχουμε δει στη σημερινή νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου ότι αρκούν επαρκούν ευρέω. Έτσι λοιπόν ε, λέμε ότι είτε δεν εμπιστευόμαστε το, η νομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου, είτε τη δεχόμαστε μάλλον, είτε δεν τη δεχόμαστε και έχουμε το σημερινό σύστημα δεν ε, ξέρουμε αν θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε τις ίδιες τις συνθήκες ή να βρούμε κάποιες παράγωγες λύσεις. Αυτό μου φαίνεται όμως ιδιαίτερα πολύπλοκο για να αντιμετωπίσουμε κάποιες περιπτώσεις που σπανιότατα θα εμφανίζονταν. Εγώ εμπιστεύομαι τους δικαστές και νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο το κύριος Ντεσούτερ. Σας παρακαλώ μη μακρηγορήστε γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θέλουμε να ακούσουμε και την απάντηση του δικαστή Τίμερμαντς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς και μόνο θα μπορούσα να πω τα εξή. Πρώτα απ' όλα κάτι πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου δεν θα είναι σε θέση ριζοσπαστικά διαφορετική, ριζικά διαφορετική μάλλον από ότι η κατάσταση άλλων συνταγματικών δικαστηρίων χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά από την προσχώρηση. Θα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν θα έχουν την ευκαιρία αυτά τα δικαστήρια, τα συνταγματικά, να εκφέρουν γνώμη. Στο Βέλιο υπάρχει αυτό το δικαστήριο, αλλά πολλές φορές οι δικαστές οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζουν κάποια θέματα δεν το πράττουν και με τον τρόπο αυτό εκτίθεται το βελικό κράτος στον κίνδυνο προτού υπάρξει μια απόφαση από το συνταγματικό του δικαστήριο, να έχει ήδη ληφθεί απόφαση από το ΕΔΑΔ. Αυτό από μόνο του δεν είναι μια ανώμαλη κατάσταση. Ο μηχανισμός προδικαστικής διαδικασίας που είναι στη διάκριση των δικαστικών αλλά δεν είναι στη διάθεση των διαδίκων των απλών των ιδιωτών περιλαμβάνει αυτό τον κίνδυνο. Αλλά σας λέω, είναι υποχρέωση για τον Εθνικό Δικαστή να θέσει ένα ερώτημα. Δεν είναι διακριτική και του ευχέρεια παραβιάζει τις υποχρέωσεις του αν απαρνείται το θέμα το προδικαστικό όταν τίθεται κάποιο θέμα ερμηνείας που είναι απαραίτητο για την έκδοση της τελικής αποφάσεως. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από ένα σύστημα θεωρώντας ότι ο Εθνικό Δικαστή δεν θα κάνει σωστά την εργασία του. Αυτό μου φαίνεται επικίνδυνη επιχειρηματολογία. Και όπω αναφέρθηκε, μία από τις δυνατότητες είναι ότι όταν ένα Εθνικός Δικαστής δεν έχει θέση ω όφιλε το προδικαστικό ερώτημα βάσει του άρθρου 276 της συνθήκης, τότε η προσφυγή που μπορεί να κάνει ο ιδιώτης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει να θεωρηθεί μη παραδεκτή για λόγους μη εξάντλησης των ενδίκων ε, μέτρων. Αλλά αυτό είναι, όπως λένε οι, αγγλόφωνες, αδικούμε κάποιον και το δέρουμε και από πάνω. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παραβίαση του άρθρου 6 τη σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα πρέπει να διαπιστώσει και το ΕΔΑ το γεγονός ότι ο Ενάγων έχει υποστεί ε, παραβίαση των δικαιωμάτων του βάσει αυτής της σύμβασης. Επίσης, η τρίτη λύση, παρά τη φαντασία της, μου φαίνεται ότι είναι επαχθής και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ενάγοντος. Οπότε θα έχουμε τέσσερις διαδικασίες σε αυτήν την περίπτωση, ενώπιον του Εθνικού Δικαστηρίου, ενώπιον του ΕΔΑΔ, έκτακτη διαδικασία που είναι κάτι ανάμεσα στην προδικαστική και την επιπαραβιάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τέταρτον που θα μπορούσε να προσθεθεί αυτό μια προσφυγή επιπαραβιάση από την Κομισιόν εναντίον του κράτους του οποίου ο Εθνικός Δικαστής αρνήθηκε να προβεί στο προδικαστικό ερώτημα. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να, να οδηγηθούμε σε μονοπάτια τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά πιστεύω. Κύριε Δικαστά, έχετε το λόγο. Κύριε μας. Μετά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Σλίτερ, από αυτές τις τόσο ισχυρές και ρωμαλαίες επιθέσεις είμαι, είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να δώσω μια, μια απάντηση. Καταρχήν για να απαντήσω στον καθηγητή Σλίτερ και για να μην υπάρξει καμία ε, σύγχυση. Εγώ δεν υποστήριξα την άποψη ότι εάν δεν υπάρξει προδικαστικό ερώτημα τότε θα πρέπει να είναι απαράδεκτη η προσφυγή από το ΕΔΑΔ. Καθε άλλο. Είπα ότι αυτή ήταν η πρώτη επιλογή την οποία μπορούσαμε να εξετάσουμε και την οποία την απέρριψα χωρίς να υπάρξει, την απέρριψα διαρρήδην. Έρχομαι λοιπόν τώρα σε αυτά που είπε ο καθηγητής Ζακέ, ο οποίος μίλησε για machine agar, δηλαδή μίλησε για ένα είδος μηχανιστικού συστήματος έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκάλ. Μήπως έχουμε μια διαδικασία η οποία γίνεται πάρα πολύ πολύπλοκη και χωρίς καμία εσωτερική συνοχή. Θα πρέπει εδώ να διαπιστώσουμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχουμε μια διπλή δυνατότητα διαδικασίας. Όταν λαμβάνεται μια απόφαση από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι μαχητή ενώπιον των θεσμικών αυτών οργάνων έναντι αυτών των θεσμικών οργάνων καλύτερα. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για προσφυγή στο ΕΔΑΔ. Αλλά αν πρόκειται για κάτι το οποίο εμπλέκει τα κράτη-μέλη, τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργεί με την αρρωγή και με την συμμετοχή των κρατών μελών. Εκεί τίθεται και το πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση, μια απλή μεταφορά του συστήματος εξάντλησης των ενδίκων μέτρων δεν θα δώσει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Γιατί είναι γεγονό ότι υπάρχουν συνταγματικά δικαστήρια που μπορεί να μην επέμβουν σε μια διαδικασία ως όφυλαν, αλλά υπάρχουν και τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών, τα οποία καταρχήν υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει καταρχήν να φτάσει κανείς εκεί να φτάσει στο, στην τελεσίδικη απόφαση προτού φτάσει στο ΕΔΑΔ. Εκεί βρίσκεται η ουσιαστική διαφορά. Γιατί ένα ιδιώτη δεν μπορεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της, το Δικαστήριο της, Ευρωπαϊκών, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλλά είναι πρόβλημα. Γιατί τελικά αυτό είναι το δικαστήριο το οποίο έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη. Δεν είναι θέμα αυτονομίας. Είναι θέμα ευθύνης του δικαστηρίου αυτού να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι παρεμβάσεων οι οποίες έχουν ασύμβατο χαρακτήρα με τα δικαιώματα αυτά από, τους, από τα άλλα θεσμικά όργανα και από τον νομοθέτη. Δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει αυτή την ευθύνη που έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και την ευθύνη που έχει. Γι' αυτό έκανα εγώ αυτή την πρόταση και βλέπω ποιες είναι οι αντιρρήσεις που διατυπώνται, αλλά όλα αυτά μου δίνουν τη δυνατότητα να διευκρινίσουμε καλύτερα τα πράγματα. Ποια ήταν η πρόταση. Η πρόταση δεν ήταν να γίνεται με μηχανιστικό τρόπο η διαδικασία. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτόματο χαρακτήρα. Και δεν πρόκειται και για διαδικασία λόγω παραβάσεως από τα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται να τροποποιήσουμε τις συνθήκες, πιστεύω ότι απλώς μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα στη συνθήκη προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΣΔΑ, γιατί είναι κομμάτι ακριβώ τη προβληματικής που εμπλέκεται από αυτή τη διαδικασία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την δυνατότητα, την προαίρεση, όχι την υποχρέωση, όταν διατυπώνει η Κομισιόν ότι υπάρχει μία προσφυγή ενώπιον του ΕΔΑΔ που αποτελεί πραγματικό πρόβλημα, βάσει του οποίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είχε την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, τότε η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει μια δήλωση, μια απόφαση υπομορφή δήλωση του, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ώστε να υπάρχει η άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βραδιπορήσει η διαδικασία κατά ανάγκη. Μπορεί να προβλέψει κανεί ένα μηχανισμό για να υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία. Υπάρχει αυτό σε άλλε περιπτώσει που εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Αυτό όμως μου φαίνεται ότι είναι μια λύση η οποία θα έχει δύο πλέον εκτήματα. Πρώτα απ' όλα λύνουμε το πρόβλημα του αποκλεισμού του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου σε ορισμένε περιπτώσει από τη διαδικασία και δεύτερον προβλέπουμε ένα ευέλικτο μηχανισμό ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι και χρονοβόρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείνουμε στο σημείο αυτό. Ξεδίσαμε όλο τον χρόνο. Ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς. Ξαναρχίζουμε στις 2. Σας είπα, έξω από την αίθουσα υπάρχει ένας μπουφές, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.